Eh, Καλημέρα Σα Θα ξεκινήσουμε αμέσω τη συνάντησή μα ε, με κάποια καθυστέρηση. Χθε είχαμε αποφασίσει ότι το 13ο θα ήταν το πρώτο το πρωί. Μετά από σχετικό έτοιμο και έγκριση του κυρίου Γκάλαγκα. Και πρόκειται για την χωρίση απαλλαγή ε, στον αφορά κοινοτικό έλεγχο αλληλεία ε, απαλλαγή 2009 σε σχέση με την υπηρεσία που θα μας παρουσιάσει σήμερα τα σχετικά και που θα παρέμβει κατά τη διάρκεια όλης της συζήτησης. Πρώτα απ' όλα κύριε Γκάρα αν συμφωνείτε να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Κώστα, τον διευθυντή της υπηρεσίας του οργανισμού, αν συμφωνείτε ή θέλετε να παρέμβετε πρώτα εσείς. Ο κύριος Κώστερ έχει τον λόγο. Καλώς ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας, έχετε τον λόγο. Thank you uh, uh, uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με την απαλλαγή για το 2009, το CFCA υπέβαλε στο Κοινοβούλιο στις 25 Νοεμβρίου την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου του 2009 από την Εσωτερική Υπηρεσία Ελέγχου της Επιτροπής που είναι επίσης και για την CFCA και ταυτόχρονα υποβάλαμε ε, μια έκθεση της CFCA για τα μέτρα που λήφθηκαν από την CFCA υπό το φως ε, των συστάσεων του Κοινοβουλίου που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα για την απαλλαγή του 2008. Επιπλέον, η βάση για την απαλλαγή είναι ε, η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Γενικά θα έλεγα ότι ε, εργαζόμαστε με την CFCA ε, στενά και με την εσωτερική υπηρεσία, υπηρεσία ελέγχου της Επιτροπής και με το ελεγκτικό συνέδριο για να βελτιστοποιήσουμε ε, τα συλλογιστικά συστήματα. Αυτό έχει γίνει από την αρχή της CFCA και έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο έχει εκπονηθεί μαζί με την εσωτερική ε, υπηρεσία ελέγχου και εφαρμόζεται από την CFCA η εσωτερική υπηρεσία ελέγχου. Ελέγχει την υλοποίηση των συστάσεων της CFCA και από τις εννέα σημαντικές συστάσεις, τέσσερις έχουν κλείσει, ε, ε, δύο ε, σημαντικές έχουν υποβαθμιστεί, δύο άλλες έχουν κρυθεί ευκτές και οι άλλες συστάσεις θα κλείσουν στο προσεχές μέλλον. Κάνοντας αυτήν την διάρθρωση, την διοικητική, ε, μοιραζόμαστε με την ΕΜΣΑ ε, ε, τον, εσωτερικό ελεγκτή, εργάζεται τρεις εβδομάδες για την ΕΜΣΑ, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας και μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την ΕΜΣΑ, η οποία υπάρχει περισσότερο από την SFCA όταν ε, χρειαζόμαστε διάφορα βοήθεια, χρειαζόμαστε πραγματογνωμοσύνη για να μπορέσουμε ε, να ε, υλοποιήσουμε διάφορες διευθετήσεις στην ε, CMCA, CFCA. Η υπηρεσία λοιπόν εσωτερικού ελέγχου είναι ικανοποιημένη με την πρόοδο την οποία έχουμε επιτελέσει και νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία τέθηκαν σχετικά με την απόδοση στο, για το 2008, οι δείκτες απόδοσης, επίδοσης, το θέμα αυτό δεν έχει κλείσει τελείως, αλλά ελπίζω ότι το 2010, για το 2010 θα κλείσει το θέμα αυτό σχετικά με την διαχείριση, την δημοσιονομική και οικονομική θα έχουμε δύσκολο χρόνο, διότι περάσαμε στο Βίγκο και ήταν δύσκολο να προβλέψουμε ε, τι θα συμβεί, ποιο προσωπικό θα έμενε ε, στην, ε, στις Βρυξέλλες, ποιο στο Βίγκο και χρειάστηκε να Επίσης να προσλάβουμε νέο προσωπικό ήταν λοιπόν δύσκολη χρονιά, όλα όμως αυτά τα προβλήματα προγραμματισμού έχουν διευθετηθεί και νομίζω ότι τα πράγματα τώρα προοδεύουν πολύ καλύτερα. Έχουμε επίπεδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού πάνω από 98%, περίπου δηλαδή 100% το 2010 δεν θα είναι το ποσοστό αυτό τόσο ψηλό, αλλά θα είναι αρκετά υψηλό παρόλα αυτά. Σχετικά με το πρόγραμμα ε, έχουμε ένα, μια καινή θέση. Η καινή θέση ε, θα πληρωθεί, ελπίζουμε, το επόμενο έτος, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι έχουμε από το establishment plan. Νομίζω ότι για τα πιο γενικά θέματα έχουμε συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών ε, και μπορώ να κάνω μερικά σχόλια πιο γενικά. Η CFCA έχει, ε, έχει μια συμφωνία έδρας η οποία ε, με την Ισπανία που επικυρώθηκε από την Ισπανία. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ ικανοποιητικό σε σχέση λοιπόν με το Βίγκο. Δεν υπάρχει ε, μια διεθνή σχολή, δεν έχουμε την κρίσιμη ε, μάζα για να μπορέσουμε να έχουμε μια διεθνή σχολή, αλλά υπάρχει μια προθυμία των τοπικών αρχών να αρχίσουν με αυτή την προσπάθεια, με, μια διεθνή σχολή, ε, γίνονται διαπραγματεύσεις. Το Βίγκο, δεν είναι το ευκολότερο μέρος για μεταφορά, για μεταφορικά μέσα. Έχουμε από το Ρίγκο στις Βρυξέλλες μία απευθείας πτήση και ελπίζουμε ότι οι περιφερειακές αρχές ε, δεν θα αφιστούν καμιάς προσπάθεια ούτω ώστε να συνεχιστεί και του χρόνου αυτή η πτήση που διευκολύνει την μεταφορά προς τις Βρυξέλλες. Σχετικά με την συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών συνεργασόμαστε με την ΕΜΣΑ, όπως είπα, την Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας και με την ΕΜΣΑ και την Frontex για επιχειρησιακά θέματα και σχετικά με την έναρξη υπηρεσιών. Ε, νομίζω έχουμε τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την χημική υπηρεσία στο Ελσίνκι. Ε, η Επιτροπή ασχολείται με όλες τις ε, διοικητικές και οικονομικές δομές και μετά ο Διευθυντής μπορεί να επικεντρώσει την προσοχή του στην βασική δραστηριότητα της κάθε υπηρεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης. Νομίζω ότι έχουμε την υποστήριξη της Επιτροπής από τις διάφορες ε, υπηρεσίες της Επιτροπής. Έχουμε πολύ καλή εμπειρία με την εσωτερική υπηρεσία ελέγχου. Άλλες υπηρεσίες βέβαια μπορούν να βελτιωθούν, πιελό. Πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός όπου δυνατόν, διότι για τις μικρές υπηρεσίες ε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πρόσθετες υπηρεσίες, ούτως ώστε το έργο των μικρών υπηρεσιών να καταστεί ευκολότερο. Σχετικά με τον συσχετισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών ε, και ε, Επιτροπής νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό. Έχουμε στην CFCA έξι μέλη της ε, Κομισιόν και έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος. Επίσης η Επιτροπή προεδρεύει και ορίζει έναν ε, πρόεδρο εκτός της Κομισιόν, ο οποίος είναι ανεξάρτητος. Νομίζω ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά και νομίζω ότι τα κράτη-μέλη είναι ικανοποιημένα με την κατάσταση και η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη. Έχουμε λοιπόν μια καλή ισορροπία, έναν καλό συσχετισμό δυνάμεων και το σύστημα αυτό δεν θα πρέπει να αλλάξει. Νομίζω ότι αυτές ήταν οι σημαντικότερες ε, παρατηρήσεις που είχα να κάνω σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κώστα. Κύριε Γκάλαγερ, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, CFCA ε, για την έκθεση και για το γεγονός ότι οι ελεγκτές και το ελεγκτικό συνέδριο έχει υποβάλει αυτή την ικανοποιητική έκθεση που μας δείχνει την κατάσταση. Η διακυβέρνηση είπατε ότι υπάρχουν έξι μέλη της Κομισιόν και ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος. Από τα 27 κράτη-μέλη ή μόνο από τα, από τα κράτη, τα θαλάσσια κράτη. Είπατε επίσης ότι έχετε υποστήριξη από την εσωτερικό έλεγχο της Κομισιόν. Υπάρχουν άλλες υπηρεσίες, είπατε, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι υπηρεσίες που θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Το 2008 υπήρξε 98% ποσοστό απορρόφησης ε, του προϋπολογισμού. Το επίπεδο εκτέλεσης Νομίζω ότι το είπατε τώρα ότι δεν θα είναι ε, τόσο ψηλή η απορρόφηση, αλλά ότι θα είναι ικανοποιητική. Γιατί δεν θα είναι τόσο ικανοποιητικό το επίπεδο απορρόφησης, το επίπεδο εκτέλεσης. Υπάρχουν δείκτες που ήταν πολύ ψηλοί το 2008 και το 2010 δεν είναι. Μήπως θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε το θέμα αυτό. Ακόμα ένα ή δύο άλλα θέματα σχετικά με τις ευθύνε και αρμοδιότητες της υπηρεσίας. Υπήρξαν ορισμένα θέματα ε, σχετικά με την Μεσόγειο θέματα κακής διαχείρισης έχει διευθετηθεί το θέμα αυτό ή υπάρχει ακόμη το πρόβλημα σχετικά μπορεί η υπηρεσία να μας επιβεβαιώσει ότι τα μέτρα ελέγχου τα οποία ε, χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα ναυτιλιακά κράτη, τα θαλάσσια κράτη έχουν πράγματι εφαρμοστεί παντού και ότι αυτοί που ε, ελέγχων στα κράτη-μέλη ε, ε, είναι ανεξάρτητα. Τι συνεργασία υπάρχει και πώς παρακολουθείτε, επιτηρείτε ότι τους ελέγχους ε, και τις ποσότητες που εκφορτώνονται κυρίως για πελαγικά είδη. Αν υπάρχει υπεραλίευση πελαγικών ειδών Νομίζω ότι αν όλες οι χώρες ε, και όλοι οι τομείς ε, μπορούν ε, να τηρήσουν τις ποσότητες αλλιευμάτων που έχουν προσδιοριστεί, τι τιμές των αλλιευμάτων θα είναι σε ρεαλιστικά επίπεδα. Ενώ αν υπάρχει παράνομη αλληλεία που εκφορτώνεται παράνομα αλλιεύματα σε οποιαδήποτε χώρα, η αξία των ε, αλλιευμάτων ε, των νομίμων και παρονόμων ε, θα είναι σε άλλο επίπεδο. Διερωτώ με αν η υπηρεσία έχει να μας πει κάτι, αν είναι ικανοποιημένη αν όλα πάνε καλά, αλλά βεβαίως οι στατιστικές των ποσοτήτων που εκφορτώνονται και οι στατιστικές ε, των εξαγωγών σε σχέση με τις ποσότητες που καταναλώνονται ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαίως αυτές οι επιβεβαιώσεις, τα στοιχεία αυτά δεν γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Χρειάζεται χρόνος για τις στατιστικές. Θέλω να ξέρω λοιπόν τι συμβαίνει με αυτήν την κατάσταση. Θέλω ε, να ε, συγχαρώ ε, την υπηρεσία και την διεύθυνση στο Βίγκο και σε κάθε ναυτιλιακό κράτος της Ευρώπης. Ξέρουμε ότι κάνετε καλά τη δουλειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Μάλιστα σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκάλαφη. Εσείς κυρία ζητήσατε τον λόγο παρακαλώ. Ε. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να σας χαιρετήσω κύριε και να σας ε, συγχαρώ θερμά. Πιστεύω ότι είναι πολύ σπάνιο από πλευράς του ελεκτικού συνεδρίου. Εγώ τουλάχιστον αυτό έζησα στη δική μου μεγάλη κοινοβουλευτική θητεία. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε τέτοιες τοποθετήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να σας συγχαρούμε θερμά για αυτό. Είπατε στα όσα μας εκθέσατε ότι το πρόγραμμα μέτρων εφαρμόστηκε πολύ καλά. Όμως δύο σημαντικά τα κλιμακώσατε και είπατε τέσσερα έχουν ε, ε, ε διευθετηθεί, δύο όχι ακόμα Ίσως αυτά τα είπατε βέβαια εσείς, αλλά θα ήθελα να μας εκθέσετε σύντομα τα σχετικά, διότι δεν κατάλαβα απόλυτα περί τίνος επρόκειτο. Και ήθελα να σας ρωτήσω επίσης όσον αφορά την παρατήρηση του κυρίου Γκάλαγκερ, πώς τους ελέγχους τώρα εσείς ε, τους βλέπετε χρηματοδοτικά υπάρχει δυνατότητα μέχρι το 2011 να τα καταφέρετε στο έργο σας ή θα υπάρξουν δυσκολίες, τι θα λέγατε. Θα ήθελα να ξέρα να μας πείτε αν ε, αυτά μπορούν έτσι να λειτουργήσουν. Κατά τα άλλα, θερμά συγχαρητήρια, κάνατε εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κώστα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Την πρώτη ερώτηση του κύριου Γκάλαχερ. Κατά πόσον το Συμβούλιο, το Διοικητικό, έχει μέλη από όλα τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ναυτιλία ή ε, περιλαμβάνονται και μέλη από άλλες χώρες. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία όμως είναι να μπορούμε να λειτουργούμε ανεξάρτητα, να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη να στηρίζεται μάλλον από τα κράτη-μέλη και να μπορεί να ασκεί του κατάλληλου ελέγχου. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της κοινή αλληλευτική πολιτικής και η Κομισιόν που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων είναι το είναι η, την αστυνόμευση θα έλεγα απέναντι τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, η υπηρεσία μας ε, χρειάζεται να είναι ανεξάρτητη και είναι τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν ε, προ τον παρόν είναι ικανοποιημένοι από τον συσχετισμό δυνάμεων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη, και η Κομισιόν, είναι ικανοποιημένα που υπάρχει ανεξαρτησία αυτού του σώματος ε, τώρα. Η υπηρεσία ε, επικουρείται από διάφορες αρχές, διάφορες υπηρεσίες ε, της Κομισιόν ε, για θέματα μισθολογίου, ασφαλίσεις, υγείας, ασθενείας. Νομίζω πως η κατάσταση εδώ μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που άπτονται του προσωπικού και χρειάζεται πρωτίστως να τα ρυθμίσουμε εμείς, θα πρέπει να υπάρχει ένα help desk στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι υπάλληλοι. Νομίζω ότι η κατάσταση λοιπόν μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Έχουμε βοήθεια επίση από την Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού έχει συσταθεί εδώ ένα help desk ε, από την ε, Γενική Διεύθυνση προκειμένου να μπορούν να απευθύνονται εκεί οι διάφορες ε, υπηρεσίες και έτσι η δουλειά να διεκπερώνεται με τρόπο πολύ πιο ευέλικτο. Έχουμε επίσης την στήριξη της Γενικής Διευθύνσης διοίκησης προσωπικού. Νομίζω πως ε, και εδώ τα πράγματα λειτουργούν αποτελεσματικά. Στο επίπεδο της ε, Διαθεσμικής Επιτροπής υπήρξε προσπάθεια να συσταθεί μια νέα υπηρεσία. Δεν ξέρω αν ε, κάτι τέτοιο θα μας βοηθούσε. Καλύτερα να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τα ισχύοντα συστήματα το 2010 και για το ποσοστό χρήσης ε, του προπολογισμού, Αυτό που έχει σημασία για το προσωπικό είναι, για το υπηρεσίες είναι το μισθή. Γνωρίζετε ότι πέρυσι είχε υπάρξει μια μείωση του συντελεστή που εφαρμόζεται στην Ισπανία. Αυτός ο συντελεστής ε, μειώθηκε κατά τη. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε μια εκτέλεση του προβλησμού λιγότερο υψηλή από την πέρυσι Φέτος ε, πρέπει να θα γύρω στο 95%. Τα πάμε λοιπόν αρκετά καλά σε φορά την εκτέλεση του προπολισμού εντός του 2010. Τώρα για τους δείκτες ε, απόδοσης ε, έχουμε ήδη τους δείκτες αυτούς για το 2009 και νομίζω ότι τα πάμε καλά. Αυτό που έχει σημασία επίσης είναι ο αντίκταπος ε, διαφόρων δράσεων σε ζητήματα συμμόρφωσης και καλύτερης συμμόρφωσης. Φροντίζουμε να υπολογίζουμε όχι μόνο την επίδοση αλλά και τον αντίκτυπο όλων των δράσεών μας ε, και το ζήτημα της συμμόρφωσης και επανέρχομαι και έρχομαι πάνω στο επόμενο ερώτημα που αφορά στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. <clears throat> Μας ε, ρωτήσατε για την Μεσόγειο. Υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα για τον ε, Ερυθρό Τόνο και συνεργαζόμεθα με τα κράτη-μέλη. <clears throat> Σας, έχω, σας έκανα ήδη ε, μια παρουσίαση την προηγούμενη φορά Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία εκρεμούν. Πάντως τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά από τότε που ξεκινήσαμε την δράση το 2008 και νομίζω πως ε, τηρήθηκαν οι ποσοστώσεις που χορηγήθηκαν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέσα τα οποία διατίθενται για τις, ε, την εξαρτήση στα κράτη-μέλη, νομίζω ότι διαθέτουμε πολλά μέσα και αυτές οι δράσεις λειτουργούν ικανοποιητικά. Από όλες τις αληθικές δραστηριότητε νομίζω ότι τουλάχιστον το ίμιση τηρήθηκαν, κάτι το οποίο είναι ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό. Δεν λέω ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, πολλά πράγματα που μένουν να γίνουν, αλλά μέρα με τη μέρα τα πράγματα βελτιώνονται και είναι πολύ καλύτερα από την προτριετία Το αυτό ισχύει για τη Βαλτική. Η Βαλτική όταν ξεκινήσαμε το 2007 οργανώσαμε μια διάσκεψη ε, εποπτείας ε, από κοινού με την ΡΑΚ για την Βαλτική συμφωνήθηκε από την Κομισιόν, ε, την ε, Αλευτική Βιομηχανία, τους επιστήμονες, την, διαδικασία, την ε, βιομηχανία μεταποίησης, ότι υπήρχε μια υπεραλίευση της τάξης του 40% Και τώρα νομίζω ότι έχουμε πλησιάσει τα επίπεδα των ΤΑΚ και η υπεραλίευση έχει μειωθεί σημαντικά στην Βαλτική. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σωστό δρόμο για την εφαρμογή αυτή ε, των απαιτήσεων συμμόρφωσης τώρα για το Βόρειο Θάλασσα. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά, η κατάσταση είναι πολύ πιο ικανοποιητική, αλλά παραμένουν κάποια προβλήματα με τα πλατή Ε, ε, σε ό,τι φορά την αλίευσή του, διότι λέγεται ότι αλίευουν ακόμα με μικρά μάτια. Τα Μπορείτε να βρείτε όλες τις ε, προφορίες στο διαδίκτυο, ότι δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας, όπως επίσης και τις παραβάσεις. Όλοι μπορούν να δουν λοιπόν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτών των κοινών προγραμμάτων. Μα ρωτήσατε για το επίπεδο ελέγχου, παραδείγματο χάρη, η υπηρεσία εργάζεται σε συγκεκριμένου τομεί και αυτοί οι τομεί αποφασίζονται από το Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενεργούμε στην ε, περιοχή ΝΑΦΟ, ΝΕΑΦΚ, αλλά και Μεσόγειο, ίσως στο μέλλον να προσταθούν και άλλες ε, περιοχές. Την τελευταία φορά όταν ε, ήμουν στην Επιτροπή Αλίας, ο κ. Στίβενσον ε, με ρώτησε σχετικά με τον ε, με το σκουμπρί. Με ρωτήσανε ποιο είναι το επίπεδο ελέγχου σε αυτές τις περιοχές. Υπάρχουν μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και αν θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει δραστηριοποίησή μας και σε άλλες περιοχές, ε, παρακαλώ να μας ενημερώσετε και θα είμαστε ευτυχείς ε, να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας ε, άμεσα και θα φροντίσουμε να επιβάλλουμε τα επίπεδα συμμόρφωσης όπως το πράξαμε με τον ερυθρό τόνο και στην Βαλτική. Και τελευταία ερώτηση σχετικά με τις συστάσεις από την ε, Εσωτερική Υπηρεσία Ελέγχου υπάρχουν μια σειρά συστάσεων και εννέα από αυτές ήταν πολύ σημαντικές. Από αυτές τις εννέα λοιπόν συστάσεις, τέσσερις πραγματοποιήθηκαν, ολοκληρώθηκαν. Μία υποβαθμίστηκε σε σημαντική και όχι πολύ σημαντική και μία υποβαθμίστηκε, υποβιβάστηκε σε επιθυμητή. Σχετίζεται, παραδείγματος με τα πρότυπα ελέγχου, μία τις συστάσεις αφορούν το σύστημα το, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να υπάρχει η λεγόμενη job description. Χρειάζεται να ολοκληρωθεί αυτή η σπάθειά μας αναφορικά με τα job descriptions ε, και το ίδιο ισχύει και για κάποια άλλα ζητήματα. που μας ε, υπέδειξε η υπηρεσία ιστορικού Αυτά. Στις εκθέσεις που στείλαμε στο Κοινοβούλιο υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ για τις πληροφορίε σας. Ε, όντως ε, ήταν αναλυτική. Κύριε Γκάλαχερ, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Η υπηρεσία απήντησε στις ερωτήσεις μία άλλη ερώτηση. Γιατί το επίπεδο εκτέλεσης το 2010 προβλέπεται ότι δεν θα είναι τόσο υψηλό όσο το 2008. Υπάρχει ίσως κάποιος λόγος γι' αυτό. Βεβαίως θέλω να συγχαρώ την υπηρεσία για το έργο το οποίο επιτελεί. Ε, νομίζω ότι επιτελεί καλή εργασία σε τομείς όπου μπορεί να υπάρχει ή υπάρχει ε, υπερβολική εκφόρτωση αλλιευμάτων, ίσως και παρανόμων. Ίσως ε, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό σε άλλη φάση σε αυτήν την Επιτροπή, διότι υπάρχουν ε, πελαγικά ψάρια τα οποία υπεραλλιεύονται. Ίσως υπάρχει υπερβολική εκφόρτωση, παράδοση τέτοιων αλλιευμάτων. Πάντως εκτιμώ το γεγονός ότι είπετε ότι θα δραστηριοποιηθείτε όπως και στην Βαλτική και όπου έχετε ε, μειώσει την υπεραλίευση σημαντικά. Και ελπίζω αυτό να συμβαίνει και σε άλλες ζώνες, σε άλλες περιοχές. Εκτιμούμε ε, αν αυτό που συμβαίνει, αυτό που ελπίζουμε ότι θα συμβεί Νομίζω ότι εν ευθέτω χρόνο θα είμαστε οι πρώτοι που θα είμαστε ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη έχουν μεγάλη ευθύνη. Εσείς δράτε ανεξάρτητα για την Επιτροπή και τις χώρες. Σας ευχαριστώ για τη σαφή σας έκθεση. Θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς κύριε Κωστέ, παρακαλώ. Ε, Όχι, γιατί... Το ποσοστό, το ποσοστό εκτέλεσης, η μισθή των υπαλλήλων υπολογίζονται και σε κάθε υπάρχει μια, ένα ποσοστό μετατροπής διαφορετικό για κάθε χώρα. Στην Ισπανία νομίζω είναι 98 και κάτι. Συνεπώς ο προγραμματισμός του προϋπολογισμού υπολογίστηκε βάσει ε, του συντελεστή μετατροπής ε, του αρχικού και αυτός ο συντελεστής μετατροπής έχει μειωθεί για την Ισπανία. Ε, συνεπώς θα έχουμε χαμηλότερο ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού, αλλά όπως είπα θα είναι ήδη πάρα πολύ ψηλό. Σχετικά με το άλλο σημείο, σχετικά με το σκουμπρί. Νομίζω ότι ο διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης DG Mare που θα έρθει νομίζω χθε στο Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό ε, ε, είχε επαφές με τον κλάδο και νομίζω ότι θα περιμένουμε ποια θα είναι η θέση της Επιτροπής αλλά αν πρέπει να ε, δραστηριοποιηθούμε επίσης ε, σε αυτή την περιοχή. Αυτό ε, νομίζω συνάδει με το πολιετές ε, πρόγραμμά μας και αν μας ζητηθεί να κάνουμε κάτι νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να φέρουμε σε πέρα σε αυτή την εργασία. Όπως είπα προηγουμένως, χρειαζόμαστε επίσης ορισμένα μέσα για να κάνουμε την εργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κώστερ. Και έτσι θα περάσουμε τώρα αμέσως στο να γνωστοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση του κυρίου Γκάλαχερ, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Παρουσίαση της γνωμοδότησης 25 Ιανουαρίου 2011, ψήφιση στην ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αλίας 15 Μαρτίου, ψήφιση στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού 28 Μαρτίου και περνάμε στην Ολομέλεια το μήνα του Μαΐου Ευχαριστώ τον κύριο Κώστερ που ήταν παρόν εδώ και ολοκληρώνεται αυτό το σημείο, το 13ο και περνάμε στο 10 της σήμερης διάταξης πρόγραμμα υποστήριξης ε, για την ενσωματωμένη πολιτική ε, θαλάσσια πολιτική. Κυρία Πατράων Νέβες, συγγήτρια. Όπως γνωρίζετε, η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Μεταφορών ζητήσαμε να είμαστε και εμείς συναρμόδιοι με βάση το άρθρο του κανονισμού μαζί με την Επιτροπή Μεταφορών από κοινού. Δεν παρίσταται η κυρία Πατραονέβες που θα της δώσω τον λόγο αμέσως. Αλλά πρώτα θα περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν συμφωνείτε πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ναι. Η κυρία Μισμαν είπατε. Εντάξει κυρία εσείς. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τον προτινόμενο κανονισμό που θεσπίζει προγράμματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενσωματωμένης ε, ε, θαλάσσιας πολιτικής υπό τις σημερινές προοπτικές για το μέλλον 2011-2012-2013. Η πρόταση κανονισμού σύμφωνα με την κανονική νομική, νομοθετική διαδικασία για απόφαση. Σημειώσαμε πολύ καλά αυτά την ε, συναρμοδιότητα της δικής σας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και τη σύνταξη γνωμοδότησης. Συγχαίρουμε την ε, συντάκτρια της γνωμοδότησης κυρία Πατράων Γιατί χρειαζόμαστε αυτόν τον κανονισμό. Πρώτα απ' όλα για να διασφαλίσουμε τη συνέχεια επειδή η προτινόμενη ρύθμιση του κανονισμού δίνει τη νομική βάση και διασφαλίζει μια αξιόπιστη και ισχυρή νομική βάση για την υποστήριξη και εκτέλεση δράσεων και μέτρων για την περαιτέρω διεύρυνση αυτών των ε, πρωτοβουλειών και δράσεων. Θέλουμε να συνεχιστούν δηλαδή οι δράσεις που έχουν αναλυφθεί και ξεκινήσει ξεκινούν και ε, συνεχίζουν ε, το πλαίσιο αυτών των προηγούμενων πρωτοβουλειών, ευθυγραμμιζόμενα πάντα όλα αυτά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου. Τελικός στόχος είναι η διασταυρούμενη ε, διαμόρφωση ενός πλαισίου μεταξύ των διαφορετικών παραμέτρων για την υλοποίηση των στόχων της Κιανής Βίβλου του 2007 του ε, κιανού εγγράφου Blue Paper και έτσι να καταλήξουμε με αυτόν τον τρόπο. Όπως γνωρίζετε, πιλωτικά προγράμματα και προκατακτικές δράσεις ε, είχαν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και που είχαν προταθεί το 2008 και μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο μέχρι τα τέλη του 2010. Χρηματοδότηση για περαιτέρω δράσεις ε, των, του IMP μέχρι το, 2000, από το, μέχρι το 2011 και 2013 δεν επαρκεί η χρηματοδότηση μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Παράλληλα, τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέτρα δεν καλύπτουν όλα τα ολοκληρωμένα μέτρα και προτεραιότητες ε, λόγω του ότι υπάρχει διασταυρούμενη ε, φύση των ε, πρωτοβουλειών αυτών. Γι' αυτό είναι αναγκαία προϋπόθεση να υπάρξει χρηματοδοτική βάση για να συνεχίσουμε. Αν δεν υπάρξει αυτός ο κανονισμός, δεν θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους ε, της θαλάσσιας πολιτικής. Η δεύτερη σημαντική αρχή που ακολουθούμε με αυτή την πρόταση είναι η αρχή της παραπληρωματικότητας, της συμπληρωματικότητας. Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότηση που προβλέπεται θα πρέπει να συμπληρώνει παραπληρωματικά υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις ε, και κονδύλια από τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες αφενός, από την άλλη πλευρά πρέπει να υποστηρίζει και να ολοκληρώνει τομεακά πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι η χρηματοδότηση δεν θα είναι επιλέξιμη για υποστήριξη από άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Προσβλέπουμε σε συνέργειες και παραπληρωματικότητα με ε, άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μορφές δράσης και κύριοι στόχοι ταυτίζονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού και εντοπίζονται εκεί. Οι προτινόμενες δράσεις θα συμπεριλαμβάνουν μελέτες, ε, πειραματικά προγράμματα και ε, δραστηριότητες, ε, φόρα από τους εμπλεκόμενους και θα συνεισφέρουν στην υλοποίηση των στόχων φυσικά των, της θαλάσσιας πολιτικής όπως αναφέρονται και στην έκθεση πρόοδου. Θα αναφέρω κάποιους από αυτούς τους στόχους. Ένας από αυτούς είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση, δεύτερον η ανάπτυξη δεξαμενών ή λεκανών, ε, θαλάσσιων λεκανών, φυσικά σε σχέση και με την κοινή αλληλευτική πολιτική. Τρίτον, η ανάπτυξη των διασταυρούμενων μέσων και εργαλείων τομεακά όσον αφορά την χρηματοδο... την, ε, το προγραμματισμό για τα μεταναστευτικά είδη ναυτιλιακές και θαλάσσιες γνώσεις και επιτήρηση. Τέταρτος στόχος είναι η προαγωγή της ε, προσέγγισης του περιβάλλοντος ε, οικολογικά των οικοτόπων. Πέμπτον, η αηφορία στην ανάπτυξη που θέλουμε να προαχθεί και όσον αφορά και την ε, απασχόληση ευθυγραμμιζόμενη με τους στόχους της στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 και θέλουμε να προαγάγουμε και τη διεθνή διάσταση όσον αφορά το IMP και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι θα είναι οι εποφελούμενοι από αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα ωφελήσει φυσικά και νομικά πρόσωπα υπό το δημόσιο και αστικό δίκαιο, οργανισμούς και υπηρεσίες, όργανα θεσμικά όργανα, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τα κράτη-μέλη και τρίτες χώρες, καθώς επίσης και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις που ακολουθούν τους στόχους της, αλληλευτικής, της θαλάσσιας πολιτικής και Τη πολιτική για την αυτιλία. Ερχόμενοι τώρα για τα δημοσιονομικά, για τα κονδύλια από πλευρά προπολογισμού. δεν έχουμε ένα καινούριο ξεχωριστό προπολογισμό, αλλά από τα διαθέσιμα περιθώρια από τον προγραμματισμό χρηματοδοτούνται και ιδιαίτερα από την κατηγορία 2 που αναφέρεται στη διατήρηση και διαχείριση των ε, φυσικών πόρων. Αυτό τι σημαίνει, ότι το περιθώριο συμπεριλαμβάνει κονδύλια που δεν έχουν κατανεμηθεί σε συγκεκριμένε ε, δράσεις για την ε, ε, πολιτική για τη θάλασσα. Έχουμε και την διαφορά όσον αφορά το περιθώριο σε σχέση με την κατηγορία 2 και τον ετήσιο προπολογισμό. Προσπαθούμε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν κονδύλια υπό την κατηγορία 2 για να χρηματοδοτηθούν οι δράσεις IMP υπό αυτόν τον προτινόμενο κανονισμό. Όπως η Επίτροπος Δαμανάκη πρόσφατα είπε στην Επιτροπή Τραν και στην Επιτροπή Αλίας ε, τέλειο Οκτωβρίου, θα καλωσορίζαμε ιδιαίτερα την υποστήριξη του Ευρωκοινοβουλίου για μια ταχεία υιοθέτηση αυτής της νομικής πράξης, αυτού του κανονισμού. Αυτό ζητήθηκε επίσης και από το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 21 Οκτωβρίου με βάση την έκθεση Μάισνερ για να ολοκληρώσω. Σημειώσαμε καλώ την υποστήριξη που εκφράστηκε από την Επιτροπή Αλληλείας στην γνωμοδότηση του κυρίου Αντινόρη που συνοδεύει την έκθεση της κυρίας Μάισνερ και ιδιαίτερα μέσα σε αυτό το πλαίσιο την, την παράγραφο 18 της γνωμοδότησης που υποστήριζε την χρηματοδότηση IMP και που προέβλεπε και υποστήριζε αυτή την συγκεκριμένη νομική πράξη, τον κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσάς, κυρία η έχετε τώρα τον λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι δεν είναι υπερβολικό να υπογραμμίζει κανείς ε, την μεγάλη σημασία που έχει η πολιτική για τα θαλάσσια θέματα και με ιδιαίτερες προσδοκίες το 2007 ξεκίνησε αυτή η ολοκληρωμένη ε, ναυτιλιακή θαλάσσια πολιτική που μέχρι σήμερα δυστυχώς ε, δεν έδωσε ακόμα τους καρπούς που αναμέναμε και προσδοκούσαμε. Υπάρχει μεγάλη προσδοκία σε σχέση με αυτή την πολιτική συνολικά και οι χώροι που είχαν δοθεί, τα, περιθώ... τα βήματα που έγιναν ήταν πολύ δειλά βήματα και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες όπως γνωρίζουμε σε επίπεδο της χρηματοδότησης, χρηματοοικονομικά. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνουμε όλο και μεγαλύτερες επενδύσεις σε αυτά τα θέματα. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια στρατηγική προσέγγιση του μέλλοντος, όχι μόνο σύμφωνα με τις αρχές μας που έχουμε προαναγγείλει στην στρατηγική 2020, αλλά σε γενικούς όρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή ανάπτυξη πρέπει να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο χερσαία επικράτεια, αλλά είναι επίσης και θαλάσσια επικράτεια και πρέπει να τοποθετηθούμε ως μεγάλη παγκόσμια δύναμη μέσα όχι στο χερσαίο πλαίσιο μόνο αλλά και στο θαλάσσιο πλαίσιο. Σε αυτό το θαλάσσιο πλαίσιο έχουμε πραγματικά ένα πεδίο δράσης πολύ διευρυμένο που αυτή τη στιγμή δεν έχει επαρκώς ε, εκμεταλλευτεί και γι' αυτό υπάρχει προσδοκία ώστε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τη θαλάσσια πολιτική με ολοκληρωμένο σφαιρικό τρόπο. Όσον αφορά το συμφέρον που η Επιτροπή Αλληλείας έχει, το ενδιαφέρον της για αυτό το πεδίο, είναι προφανές το ενδιαφέρον αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι η ολοκληρωμένη ναυτική πολιτική, θαλάσσια πολιτική θα πρέπει να έχει μια ολιστική προσέγγιση, οριζόντια, εγκάρσια, με όλες τις δραστηριότητε, με κοινωνικό πλαίσιο, περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο πλαίσιο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας σε όλους τους, σε όλα τα πεδία της κοινωνικής δράσης και δραστηριότητας και πιστεύουμε πραγματικά ότι είναι δυνατό μέσα στις διαφορετικές δράσεις να καλύψουμε κάθε έναν από τους ε, τομείς αυτούς. Κάθε τομέα θα υποφεληθεί αν έχουμε μια σφαιρική, αρθρωμένη, σύνθετη πολιτική. Και έτσι και ο τομέας της επίσης. Ο τομέα της μπορεί και πρέπει να προσεγγίζεται από μια ολοκληρωμένη ναυτική και θαλάσσια πολιτική που πραγματικά τον τομέα της αλληλεία θα τον θεωρεί έναν από τους πιο ζωντανού και θεμελιώδεις μέσα στα πλαίσια των δράσεών μα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο με μεγάλη εκτίμηση βλέπουμε πρώτα απ' όλα όπω αναφέρθηκε τα δειλά βήματα που έγιναν μέσα σε αυτό το ε, το σε αυτό το πλαίσιο και αυτά που είναι οι χρηματοδοτικές προσδοκίες ε, για, αυτό τον, ε, για αυτή τη μεταβατική περίοδο μεταξύ 2011-2013 Πραγματικά αυτό είναι εδώ το οποίο διακυβεύεται, το οποίο τίθεται ε, επί τραπέζης. και από τα ε, λόγια και τα σχόλια που άκουσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκλίνουν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή είναι να ξέρουμε αν θα έχουμε την χρηματοδοτική υποστήριξη που είναι αναγκαία για να καταφέρουμε να συνεχίσουμε τα πιλωτικά προγράμματα που βρίσκονται υπό εξέλιξη και πραγματικά να δώσουμε συνέχεια συνέχεια στα δειλά βήματα που έγιναν όσον αφορά τη θαλάσσια πολιτική με προοπτική και προσδοκία να καταφέρουμε να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα το 2011 και καθοριστικά πλέον το 2013, ώστε να καταλήξουμε σε μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρώπης μέσα στο πλαίσιο που σκιαγράφησα πιο πριν, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι η Ευρώπη δηλαδή πρέπει να κερδίσει αυτό τον αγώνα, αυτή τη μάχη του ανταγωνισμού που δίνει για την παρουσία της στην παγκόσμια σκηνή, όχι μόνο στην χερσαία επικράτεια, ε, στην ε, ε, γεωγραφία της χερσαίας επικράτειας αλλά και στη θάλασσα. Έχουμε κύριο μεγάλο ενδιαφέρον στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και θα πρέπει πολύ προσεκτικά να στρέψουμε το βλέμμα όχι μόνο για αυτή την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική αλλά και για το πώς ε, τα θέματα αλληλείας θα έχουν το πλαίσιο που τους αξίζουν μέσα σε αυτή την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και θα παρακολουθήσουμε και θα συνοδέψουμε όλες αυτές τις διαδικασίες ασκώντας τη μέγιστη πίεση ώστε τα χρηματοοικονομικά μέσα να διατεθούν και να διασφαλιστούν όπως πρέπει και θα πρέπει επιτόπου να προαχθούν όλες οι νέες ιδέες και προτάσεις που έχουν υποβληθεί και που προσυπογράφουμε να εκτελεστούν με το σωστό τρόπο και συγκεκριμένα εξειδικευμένο, χειροπιαστό τρόπο όπως προσδοκούμε και αναμένουμε και ουσιαστικά ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί και που έχουν παρουσιαστεί. Επ' αυτόν κυρίως είχα να πω ε, να κάνω τα σχόλιά μου. Δεν έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όσον αφορά την χρηματοδότηση, ελπίζω ότι, ε, πιστεύω ότι ήδη αναφέρθηκε ότι πρέπει να σημειωθεί πρόοδος να διασφαλιστούν τα κονδύλια και πιστεύω ότι πραγματικά εδώ θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πατράου Νέβες. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις να διατυπώσω στην Επιτροπή σχετικά. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι το Συμβούλιο, στο Συμβούλιο υπάρχουν προβλήματα με αυτή την πρόταση από ό,τι ακούω. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε ακριβώς πού βρίσκονται αυτά τα προβλήματα. Ένα πρόβλημα νομικής βάσης ίσως επίσης. Και πραγματικά θα ήθελα να γνωρίζω ποιο είναι το πρόβλημα της νομικής βάσης. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της επιτροπολογίας, πάλι θα ήθελα να γνωρίζω σε σχέση με τη συζήτηση τι γίνεται. Εσείς προτείνετε μια συμβουλευτική επιτροπή. Τα κράτη-μέλη προτείνουν μια κανονιστική, ρυθμιστική επιτροπή. Θα ήθελα να ξέρω γιατί προτιμούν ρύθμιση και κανονιστική, κανονιστικά πλαίσια τα κράτη-μέλη, ενώ εσείς προτείνετε μια συμβουλευτική επιτροπή. Και το θέμα της χρηματοδότησης. Για τη χρηματοδότηση πάλι υπάρχουν προβλήματα στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα ουσιώδη προβλήματα. Το ποσό, τα ποσά ε, που προτείνονται είναι αυτά τα οποία εσείς προτείνετε να συμπεριληφθούν στην κατηγορία 2 ή στο περιθώριο της κατηγορίας 2. Εγώ προσωπικά έχω κάποιες αμφιβολίες γι' αυτό και θα το ξαναθέσω το θέμα αν μπορεί να ενταχθεί αυτό στην κατηγορία 2 ή όχι. Έχω αμφιβολίες εγώ. Θα ήθελα να μας αποσαφηνίσετε όμως γιατί είναι σκόπιμο να βρίσκεται στην κατηγορία 2 και όχι σε άλλη κατηγορία η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡ είναι στην κατηγορία 2 και σε σχέση με την αλληλεία θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι το περιθώριο της κατηγορίας 2 θα είναι διαθέσιμο, δηλαδή για τα κονδύλια για την αλληλεία. Θα ήθελα να μας αποσαφηνίσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Και γι' αυτό θα σας δώσω χωρίς ε, ε, να χρονοτριβώ τον λόγο. Α, υπάρχει κι άλλο σημαντικό θέμα εδώ. Πιστεύω ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σχετίζεται με το θέμα της έρευνας, αλλά ιδίως στην επικέντρωση την οικοσυστημική των οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος. Δεν υπάρχουν όμως κονδύλια και δεν έχει αναφερθεί αυτό. Θα ήθελα να ξέρω από εσά πότε θα προβλέψετε, πώς θα προβλέψετε αυτή η ολοκληρωμένη πολιτική για τη θάλασσα να μπορέσει να λειτουργήσει και να υπάρχει μια πραγματικά πάγια και ισχυρή επιστημονική βάση για να μπορούν όλα αυτά να λειτουργήσουν σωστά. Όλες αυτές τις ερωτήσεις μπορείτε να τις απαντήσετε τώρα παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσουμε την ερώτηση που αφορά στον προπολισμό. Μιλάμε για τον παρελθόν. Στο παρελθόν τα προγράμματα ήδη χρηματοδοτούνται από τα περιθώρια του κεφαλαίου 1. Του κεφαλαίου 2, συγγνώμη. Αυτό είναι ένα στοιχείο συνέχειας, ότι δηλαδή για τη νέα ε, δημοσιονομική περίοδο περίοδο ε, 2013 τα χρήματα θα προέρχονται από αυτό το συγκεκριμένο κεφάλαιο, ιδιαίτερα σε φορά την ε, διατήρηση και τη διαχείριση των ε, εθνικών πόρων. αυτό έχει καταδειχθεί ότι είναι το καταλληλότερο κεφάλαιο για την ε, χρηματοδότηση της ολοκληρωμένης θαλάσσης πολιτικής. Τώρα, για το ζήτημα των Συμβουλίων και των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται εκεί. Δεν είμαι σε θέση να μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με τις εν λόγω συζητήσεις. Σε ό,τι αφορά τη νομική βάση, να σας πω ότι υπάρχει πρόβλημα για την νομική βάση, διότι υπάρχουν πολλαπλές νομικές βάσεις για αυτόν τον κανονισμό και αυτό οφείλεται στους πολλαπλούς στόχους ε, της ε, πολιτικής ε, και των εγκάρσιων ζητημάτων. Υπάρχουν τα άρθρα 4, 4 και 77, 2 που αφορούν στο άρθρο το σχετικό άρθρο της ε, συνθήκης, το Συμβούλιο ε, πρότεινε να διαγραφούν οι δύο αυτές τις αναφορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα δούμε επίσης ποια θα είναι και η στάση του Κοινοβουλίου. Τώρα για τις συμβουλευτικές επιτροπές η Κομισιόν πρότεινε αυτή την επιτροπή, διότι θεωρούμε ότι είναι το καταλληλότερο φόρουμ για αυτά τα χαμηλά ποσά. Εδώ μιλάμε για 50 εκατομμύρια ευρώ που είναι ένα πολύ μικρό, πολύ χαμηλό ποσό. Δεν έχει πολλές ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις για τα κράτη-μέλη που θα χρειαζόταν μια κανονιστική επιτροπή τώρα. Το ζήτημα της επιτροπολογίας φυσικά άπτεται της νέας διαδικασίας. Ε, αυτό θα το δούμε και θα σας αναφέρουμε σχετικά όταν θα έχουμε προοδεύσει στον κομμάτι αυτό. Τώρα, αναφορικά με την έρευνα, ο κανονισμός ε, προβλέπει δράσεις για τα θέματα γνώσεων στον θαλάσσιο τομέα και συλλογή στοιχείων για ένα ποσό 22 εκατομμυρίων πάνω κάτω. Είναι ενδεικτικό το ποσό αυτό, διότι τα ποσά συμπεριληφθούν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Τώρα, η θαλάσσια και η θαλάσσια έρευνα ε, προβλέπεται και από άλλα προγράμματα όπως το 7ο πρόγραμμα που προβλέπει την κοινή πρωτοβουλία για τους ωκεανούς που ξεκίνησε φέτος το καλοκαίρι και υποστηρίζει την θαλάσσια και ναυτική έρευνα. Εδώ έχουμε τη σημαντικότητα των δράσεων, έχουμε την Γενική Διεύθυνση RTD και αφετέρου έχουμε και τις δράσεις για τις γνώσεις, τις δεξιότητες. θαλάσσια έρευνα που περιέχεται στην, ε, στην ε, οδηγία για την 2020. Ε, Ελπίζω να μπορέσει να καλυφθεί διότι αυτό θα ήταν κακό. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ πιστεύω ότι το θέμα της έρευνας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν υπάρχει αυτό, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική δεν θα είναι επιτυχία. Και γι' αυτό τώρα, κυρία Ισηγήτρια, όσον αφορά για την ε, χρηματοδότηση, για την ε, έρευνα, για την ε, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, πρέπει να διασφαλιστεί αυτή. Διαφορετικά θα κάνουμε ένα λόγο για ένα θέμα, όπως μέσα στο πλαίσιο της αλληλείας για την επιστημονική έρευνα που δεν θα έχει χρηματοδότηση. Επιμένω, το θέμα της χρηματοδότησης θα πρέπει να τεθεί σε βάθος στην κατηγορία 2 θα ενταχθεί ή αυτό το θέμα είναι θεμελιωδός θέμα μεταφορών ή τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου σχετικά και πιστεύω ότι πρέπει να μελετήσουμε το θέμα της χρηματοδότησης και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο αφορά ακριβώς ε, το θέμα ε, της ε, χρηματοδότησης υπό το δικό μας πρίσμα σε σχέση με την Επιτροπή Μεταφορών. Προφανώς μέσα στο πλαίσιο της κατηγορίας 2, αν λοιπόν σε σχέση με την Επιτροπή Μεταφορών, αυτή θα είναι η Επιτροπή αρμόδια για το μέλλον για αυτό το θέμα, να είναι αυτό σαφές. Εγώ πιστεύω ότι θα δώσουμε μάχη για αυτό το θέμα διότι εμείς εδώ πρέπει να έχουμε σαφείς ε, γραμμές ε, αρμοδιοτήτων για τα θέματα μας. Λοιπόν, τούτου λεχθέντος, η κυρία Πατράου, για να ολοκληρώσει παρακαλώ, έχει τον λόγο. Πολύ ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ τα θέματα στα οποία επικεντρωθήκατε και κυρίως όσον αφορά τα θέματα έρευνας. Είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη όσον αφορά την ανάγκη που υπάρχει να διασφαλίζουμε μια προσέγγιση των ωκεανών στο ευρύτερο πλαίσιο και σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συστημικά, οικοσυστημικά να έχουμε μια σωστή προσέγγιση. Για τα θέματα αλίας αρκετές φορές υπήρξαν αμφιβολίες ε, όσον αφορά την τομεακή συλλογή και συγκρότηση στοιχείων. Αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά είναι μια ολοκληρωμένη κάποια μορφή ή τρόπος ε, έρευνας που θα επικεντρώνει όλα τα στοιχεία κεντρικά και θα μπορεί να δημιουργεί συνθετικά ένα ολοκληρωμένο όραμα, μια συνολική προσέγγιση των ωκεανολογικών θεμάτων και των ωκεανών. Αν δεν γίνει αυτό θα συνεχίσουμε να έχουμε μόνο τομεακές δράσεις, περιορισμένες δράσεις, χωρίς, συνολικές ε, επιπτω... Ε, χωρίς συνολική μελέτη επιπτώσεων. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πτυχή γι' αυτό. Και εφόσον δεν θα υπάρχει αυτή η γενική προσέγγιση για τους ωκεανούς και τις θάλασσες, θάλασσες η ολοκληρωμένη ε, πολιτική για τη θάλασσα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Και το θέμα της χρηματοδότησης είναι σημαντικό διότι πραγματικά υπήρξαν μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά αυτή την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και βλέπουμε ότι δεν προχωρεί σύμφωνα με τις προσδοκίες ε, και τις ελπίδες μας ε, για τα χρηματοοικονομικά θέματα. Και για άλλη μια φορά αυτή η πρόταση ε, του κανονισμού για θέματα χρηματοδοτικά βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ή των ε, αντιπαραθέσεων. Λοιπόν, σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν εδώ, αυτά είχαν από κυρίως πρέπει να δούμε από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν η δέσμευση για αυτή την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο επίπεδο αυτό που παρουσιάστηκε το 2007 διατηρείται σήμερα ή όχι. Και μπορούμε να αξιολογήσουμε αν διατηρείται ή όχι αυτό το επίπεδο μόνο αν υπάρξουν συγκεκριμένες εξειδικευμένες προσπάθειες και προτάσεις για να δοθεί συνέχεια σε αυτό που ξεκίνησε το 2007 και να μην σταματήσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επιτροπή. Ολοκληρώθηκε το σημείο 11. Στην επόμενη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί η συγκήτρια το, η έκθεση και θα καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι το 12 και που είναι για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Μαρόκου για την ε, ε, ρύθμιση των θεμάτων των αγροτικών γεωργικών προϊόντων που εισηγητής γι' αυτό είναι ο κύριος Ρωμέβα. Η Επιτροπή είναι, ίντα είναι η αρμόδια της ουσίας για αυτό το θέμα. Η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή συντάσσει γνωμοδότηση θα ήθελα να δώσω τον λόγο αμέσως στον κύριο Ρωμέβα, πιο πριν πρωτού δώσω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε τον λόγο κύριε Ρωμέβα. Σας ευχαριστώ πολύ γοργά πρόεδρε, επειδή πρέπει να ακούσουμε και τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν πάση περιπτώσει, δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις θα είχα να διατυπώσω για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε κάποιες απαντήσεις σήμερα το πρωί. πρώτη, ήδη την υπενήχθηκα εχθές, αφορά το γεγονός ότι όλοι μας είμαστε, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή είναι μια έκθεση που δεν είναι μόνο τεχνικού χαρακτήρα. Υπάρχει μια πολιτική συνιστόσα που είναι, μας κάνει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Είναι σημαντικό να είναι σαφή τα πράγματα για αυτά τα θέματα. Αυτή τη στιγμή έρχομαι για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όπου γίνεται παρουσίαση και των εκπροσώπων της Πολυσάριο, της Δυτικής Σαχάρας και ε, σε σχέση με τους εκπροσώπους του Μαρόκου Λοιπόν, το πλαίσιο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Δεύτερον, υπάρχει μια νομική πτυχή, διεθνής νομική πτυχή, που και γι' αυτό πρέπει να έχουμε ευαισθητοποιηθεί και να είμαστε ιδιαίτερα υπεύθυνοι όταν έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Και με άλλες αφορμέ είχαμε παρόμοιε συζητήσει και σε σχέση και με τη Συμφωνία Λίας που παρότι δεν είναι το ίδιο, κάπως συσχετίζεται και εγώ συντάκτης γνωμοδότησης κάνω τους εξή ε, ε, τις εξής σκέψεις. Πρώτα απ' όλα, με σαφή τρόπο θα ήθελα να ξέρουμε ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την νομική αξιολόγηση της νομικής ε, πτυχής της Συμφωνίας Αλίας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να κατανοήσουμε προς ποια κατεύθυνση πορευόμαστε και τι συμβαίνει. Δεύτερον, θα ήθελα επίσης να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει με το συγκεκριμένο κείμενο που έχουμε μπροστά μας και εξετάζουμε ποιο μέρος των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αλληλείας προέρχονται από την επικράτεια της Δυτικής Σαχάρας. Διότι αυτό αφορά και τη νομική βάση αυτής της συμφωνίας. Και τρίτον, ακολουθώντας ε, τη θέση του εισηγητή στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή επί της ουσίας ε, την ΙΝΤΑ, που είναι ο Ζωζέ Μποβέ, και που ζήτησε να υπάρξει γνωμοδότηση νομική από τις νομικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση αυτής της συμφωνίας, μια και εμείς ως ε, Επιτροπή Αλληλείας γνωμοδοτούμε, πρέπει να αναμείνουμε να υπάρξει αυτή η νομική γνωμοδότηση εσωτερικά, να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο και η νομική βάση επί της οποίας μπορούμε να κινηθούμε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να γνωμοδοτήσουμε εμείς. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πραγματικά ποια είναι η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το κείμενο. Ποιες είναι οι προτάσεις ε, που ε, πρέπει να εξεταστούν και τι γίνεται και τι προβλέπετε, ιδιαίτερα όσον αφορά με την νομική βάση και ποια θα είναι η εφαρμογή σχετικά των ε, συμφωνιών που αφορούν και κατεχόμενα εδάφη όπως αυτό της Δυτικής Σαχάρας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι το ζήτημα της Αλίας δεν εξετάζεται εδώ, δεν υπάρχει κάποιος πρόσωπος σχετικά. Υπάρχει εκπρόσωπο από τη Γενική Εύση Μάρα για να μας μιλήσει για τη Συμφωνία Σύνδεσης και για τα γεωργικά προϊόντα και ελευτικά προϊόντα. Δώσε το λόγο στον κύριο Βαν Ρέικ. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή για τις παρατηρήσεις του και τα θέματα τα οποία παρουσίασε και ανέφερε. Βεβαίως υπάρχει σημαντική διεθνής διάσταση σε αυτή τη συμφωνία σχετικά με τις, τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό το πλαίσιο το διεθνές προέρχεται από τη συμφωνία Euromed που υπογράφηκε το 1996 και τέθηκε σε ισχύ το έτος 2000, όπως γνωρίζετε ασφαλώς, όσον αφορά το αλλιευτικό μέρος αυτής της συμφωνίας, το 2000 υλοποιήθηκε η πλήρης απελευθέρωση της εμπορίας αλλιευμάτων σχετικά με τις εισαγωγές από το Μαρόκο. Όλες οι εισαγωγές από το Μαρόκο μπορούσαν να εισέλθουν δωρεάν, αδασμολόγητα ε, στην, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάγει προϊόντα. Λάβαμε την εντολή το 2005 για να επαναδιαπραγματευτούμε αυτή την συμφωνία, να βελτιώσουμε περαιτέρω κατά κάποιο τρόπο τις εμπορικές συνθήκες και βεβαίως για το τμήμα το, ε, των αλλιευμάτων βασικός μας στόχος ήταν να εξισορροπήσουμε αυτή την κατάσταση ε, και να επιτύχουμε πλήρη απελευθέρωση για ε, τις δυνητικές μας εξαγωγές στο Μαρόκο επιτύχαμε αυτό το στόχο. Η μεγάλη πλειονότητα των εξαγωγών, κυρίως ε, γαρίδες, ε, θα απελευθερωθούν πλήρως ε, αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ αυτής της συμφωνίας σχετικά με τα άλλα προϊόντα σε 5 ή 10 χρόνια θα επιτευχθεί η πλήρης απελευθέρωση. Και πάλι εδώ, εφόσον βρίσκομαι στην Επιτροπή Αλίας, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας πάνω σε αυτό το απλό γεγονός. Τώρα, με αυτό το, στη συμφωνία που έχουμε επιτάπητος, δεν παρέχουμε νέες παραχωρήσεις στο Μαρόκο. Αντιθέτως, είναι τώρα η δική μας σειρά να ωφεληθούμε από τη συμφωνία και ε, χαίρομαι που μπορώ να επισημάνω ότι θα επιτευχθεί η πλήρης απελευθέρωση και για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, οι οποίες μέχρι τώρα ήταν δασμολογημένες. Σχετικά με την προέλευση των προϊόντων, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είχαμε σκληρές διαπραγματεύσεις ε, σχετικά με τους κανόνες προόλευσης ε, που θα ισχύσουν για αυτή τη συμφωνία από μαροκινής πλευράς υπήρξε ε, ένα αίτημα να υπάρξει κάποια χαλάρωση στους αυστηρούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την χώρα προέλευσης, αλλά αντισταθήκαμε και οι κανόνες σχετικά με την προέλευση θα ισχύσουν και στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες προέλευσης θα εξαρτώνται από την σημαία των πλοίων που αλλιεύουν σε αυτή την περιοχή. Μια σύντομη πληροφορία σχετικά με το στάδιο έγκρισης αυτής της συμφωνίας. Εάν όλα προχωρήσουν ικανοποιητικά, τότε θα εγκριθεί η απόφαση που θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να υπογράψει τη συμφωνία. Αυτή η άδεια για την υπογραφή θα υιοθετηθεί ως, θέμα όχι προς συζήτηση στις αρχές του Δεκεμβρίου και η συμφωνία θα μπορέσει να υπογραφεί από τα δύο μέρη στο περιθώριο ε, του Συμβουλίου Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου στα μέσα του Δεκεμβρίου και μετά θα επανέλθουμε σε εσά με αυτήν την πρόταση που έχουμε επιτάπητος και θα ζητήσουμε την έγκριση των, ε, της συμφωνίας των συμπερασμάτων της συμφωνίας. Αυτά έχω να σας πω ως Γενική Διεύθυνση Εμπορίου για το εμπορικό τμήμα της συμφωνίας και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ράμπο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος εφόσον ο κύριος Σόμοβη ανέφερε σαφώς ότι το καθεστώς που συμφωνήθηκε βασιζόταν σε μια αρχή, δηλαδή την προέλευση του προϊόντος, η προέλευση του ε, προϊόντος ε, η εθνικότητα του προϊόντος εξαρτάται από το αλλιευτικό πλοίο, από τη σημαία του αλλιευτικού πλοίου που αλλιεύει αυτό το προϊόν. Τα προϊόντα ε, που καλύπτονται είναι μαροκινά προϊόντα και ευρωπαϊκά προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα που αλλιεύονται από σημαία ευρωπαϊκή ή ε, με σημαία μαροκινή. Αυτή είναι η κατάσταση για την ώρα και έτσι αντιμετωπίζονται τα αλλιευτικά προϊόντα, έτσι όπως συμφωνήθηκε στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Νομίζω πως ο κύριος Ρωμέβα δεν ικανοποιήθηκε. Θα ήθελα κάποια μέρα να συζητήσουμε σοβαρά το ζήτημα του κανόνα προέλευσης Γνωρίζω πως ε, το ζήτημα αυτό ε, συζητείται από τρίτες χώρες ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γενική Διεύθυνση Trade έχει, γενική, έχει μια άποψη διαφορετική από την Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Εμείς λοιπόν ως Επιτροπή Αλίας θεωρώ ότι δεν μπορούμε να επισερχόμαστε σε συμβιβασμούς, τη φιλελευθερωποίηση, τη ενισχύσεις προς τρίτες χώρες και να μην λαμβάνουν υπόψη τα ευαίσθητα προϊόντα, την ευρωπαϊκή βιομηχανία, τον ευρωπαϊκό κλάδο αλληλεία κλπ. Κατά την άποψή μου λοιπόν τα θέματα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Νομίζω πως το παράδειγμα της Νέας Γουινέας ε, μας ε, δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα και ξέρουμε πίσω ότι πολλές φορές είναι θέματα τα οποία επηρεάζουν και τις τρίτες χώρες και τον αλληλευτικό κλάδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν κάποια μέρα να μπορέσουμε να έχουμε μια γενικότερη και ειλικρινή συζήτηση με τη Γενική Διευθυνσή Τρέιντ και Γενική Μάρε προκειμένου να δούμε προς τα που πηγαίνουμε και τι πιθανότητες υπάρχουν να εφαρμοστεί μια κοινή στρατηγική από όλους τους εμπλεκόμενους, διότι βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος. Ε, θέλετε να θέσετε περαιτέρω ερωτήσει, έχετε το λόγο κύριε Ρωμουέδα. Θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία και σε άλλους συναδέλφους που θέλουν να παρεύουν. Διακόπτη Πρόεδρος. Ναι, ας λάβουμε το λόγο και κύριος Κάντεκ. Μια από ο κύριος Ρωμέδα θέλει να λάβει το λόγο πριν από αυτόν, θα το πράξω προκειμένου για τις συμφωνίες Αλίας με το Μαρόκο. Πρόκειται για μια συμφωνία που νομίζω ότι ε, ε, λήγει στην 23η Φεβρουαρίου. Άρα λοιπόν ε, οι Μαροκινοί ανησυχούν και θέλουν να γνωρίζουν κατά πόσον θα ανανεωθεί αυτή η συμφωνία ή όχι. Έχουν ζητηθεί κάποιε πληροφορίε από την Κομισιόν και από ό,τι γνωρίζω οι μαροκινοι ανησυχουν και θελουν να γνωριζουν κατα ποσον θα ανανεωθει αυτη η συμφωνια η οχι εχουν ζητηθει καποιες πληροφοριε απο την κομισιον και απο οτι γνωριζω μαροκινές αρχές ε, υπέβαλαν στην Κομισιόν τα απαραίτητα έγγραφα, τουλάχιστον αυτά που τους είχαν ζητηθεί, έτσι μου είπαν τουλάχιστον οι Μαροκινοί, ιδιαίτερα το θέμα που άπτεται των κλαδικών ενισχύσεων, κατά πόσον κατανέμονται σωστά στο σύνολο της Μαροκινής εντός εισαγωγικών επικράτειας. Φαίνεται πως σύμφωνα με τις προφορίες που λάβαμε, ότι τομεακή βοήθεια κατανέμεται σωστά στο σύνολο της παράκτιας επικράτειας Σούμα Ρόκου από την Ταγκέρνη με το Μαλιμπού. Διότι εδώ έγκυται το ζήτημα. Πρόκειται για ένα καθαρά πολιτικό θέμα. Το ξέρουμε πολύ καλά. Διότι υπάρχει το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας και των Πολυσάριων. Εδώ βρίσκεται λοιπόν το πρόβλημα. Φυσικά αυτό δεν εξαρτάται από την Επιτροπή μας, αλλά γνωρίζω πως χθε ε, το μέτωπο Πολυσάριο συζήτησε με την Κομισιόν στις Βρυξέλλες και το Μαρόκο θα συζητήσει σήμερα εντός 40 λεπτών στις 11 η ώρα σχετικά με αυτήν την πολιτική κατάσταση που επικρατεί σε αυτόν τον τομέα του Μαγκρέμπα. Λυπούμεθα που ο τρίτο εταίρος δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση, την Αλγερία δηλαδή, που έχει και αυτή θέση στην όλη συζήτηση σε ό,τι με αφορά. Πιστεύω πως θα ήταν παρακεντρευμένο φαινό για την τοπική πολιτική ισορροπία αλλά και για την ευρωπαϊκή αλία η συμφωνία αυτή να μην ανανεωθεί ή να μην τύχει επαναδιαπραγμάτευσης φόσον οι ενισχύσεις κατανέμονται δίκαια και στη Δυτική Σαχάρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, ανανεωθεί η συμφωνία, διότι όλοι θα την πληρώσουν, οι Μαροκινοί, οι κάτοικοι της Σαχάρας και οι Ευρωπαίοι. Αυτά είχα να σας πω σήμερα, να φάει και να ακολουθούμε εκ του σύνεγγης, διότι το θέμα είναι κατεπίγον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Άντρες Μπαρέα, ευχαριστώ πρόεδρε. Λοιπόν, αληθεύει ότι οι διεθνείς συμφωνίες έχουν μια πολιτική συνιστόσα. Γιατί γι' αυτό συνάπτονται οι διεθνείς συμφωνίες. Βρισκόμαστε εδώ όλες τις μέρες και σε άλλες κοινοβουλευτικέ επιτροπές όπως την ΙΝΤΑ κάνοντας λόγο για διεθνείς συμφωνίες με χώρες που θέλουμε να βοηθήσουμε να αναπτυχθούν. Και γι' αυτό είναι θεμελιώδες να διατηρηθούν αυτές οι διεθνείς συμφωνίες υπό αυτό το πρίσμα. Είναι καλό αυτό να δίνουμε βοήθεια, να σύνδρομη για την ανάπτυξή τους σε αυτές τις χώρες, εμπορικά και τα λοιπά. Τι γίνεται με το Μαρόκο. Κάνοντας λόγο υπό το πρίσμα το εμπορικό, όπου στην Επιτροπή Αλίας μας αφορά η Συμφωνία Αλίας ή στην Επιτροπή Γεωργίας η Συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα, είναι ένα θέμα αυτό. Αν κάνουμε λόγο για τη νομική πτυχή και τα προβλήματα της Δυτικής Σαχάρας, νομίζω ξεπερνούν τα πλαίσια αυτής της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Το έχουμε επαναλάβει αυτό επανειλημμένα σε αυτή την Επιτροπή. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε κυρίω σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή να επιλύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο 30 χρόνια εκρεμεί και δεν έχει επιλυθεί. Και εδώ θα πρέπει να φυσικά ζητείτε να επιληθεί, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό μέσα στους κόλπους της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Δεν μπορεί εδώ να επιληθεί. Σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, σε αυτή την έκθεση γνωμοδότησης πρέπει να δούμε την συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα αφενός, την συμφωνία για τα αλληλευτικά προϊόντα για την αλληλεία αφετέρου, για την αλληλευτική συμφωνία. Εδώ, σε σχέση με την ε, ίδια την μεικτή επιτροπή και εδώ διεκδικούμε το, τα θέματα της ε, ε, μεικτής επιτροπής που φαίνεται ότι αγνοείται σε αυτό το θέμα θα πρέπει να, να αναλυθεί εκείνη το ανέλησε και τα παρουσίασε αν αυτό αφορά τον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας και αν όχι να ληφθεί αυτό υπόψη. Αν όμως αφορά αυτή την περίπτωση τότε να τεθεί στο τραπέζι και να μπορούμε να δούμε περί τίνος πρόκειται. Κάτι το οποίο εκρεμεί. Κάποιοι λένε έχει συμβεί, κάποιοι άλλοι όχι, λένε ότι όχι δεν γίνεται, δεν, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θέλουμε να έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας, είναι θεμελιώδες. Υπό το γεωργικό πρίσμα φαίνεται ότι η Επιτροπή Γεωργίας δεν είχε κανένα πρόβλημα. Αν αυτό είναι το θέμα για την αρμοδιότητα των παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ τίθεται ένα πρόβλημα. Και αυτό είναι η τροποποίηση του κανονισμού μέσα στο ε, πλαίσιο εισαγωγή αυτών των προϊόντων. Εμεί στην Επιτροπή Αναφορών ζητήσαμε να τροποποιηθεί αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο θέμα απόλυτα τελείω διαφορετικό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι εδώ, αν εξετάζοντα τι εμπορικέ συμφωνίε, ε, εμπορικέ υπό το πρίσμα της γεωργίας με σύνταξη έκθεσης νομοδόσης ή για τη Συμφωνία Αλίας, αυτό πρέπει να δούμε είναι αν υλοποιείται αυτή η Συμφωνία για το Εμπόριο από τις μικτές επιτροπές. Αν εξειδικευμένα ε, ε, υλοποιείται και υπάρχει συμμόρφωση ή αν υπάρχει κάποια τροποποίηση. Μέσα σε, αυτή, σε αυτό το αδιέξοδο βρισκόμαστε λόγω εξωτερικών παραγόντων και λόγων και πρέπει να επιληθεί αυτό και πρέπει υποχρεωτικά να επιληθεί αλλά δεν είναι μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής που μπορούν να επιληθούν όλα αυτά τα θέματα. Eh, Ευχαριστώ κύριο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εάν ε, να μιλήσουμε για αλληλεία, δεν έχουμε να προσθέσουμε πολλά πάνω στο ζήτημα. Θεωρώ πως ε, όταν μιλάμε για αλληλεία και αλληλευτικά προϊόντα, Ε, είναι ένα κομμάτι τη όλη συζήτηση, διότι το βασικό είναι τα γεωργικά προϊόντα. Μπορούμε να μπλάμε για συμφωνία αλλίας αν θέλετε, αλλά δεν είναι το αντικείμενο αυτή τη συμφωνία. Εντάξει, υπάρχουν πολλά θέματα που οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, έχουμε τι θέσει μα, υπάρχει το ζήτημα τη πρόέλευση των προϊόντων, αλλά και οι διατάξει οι υγειονομικέ και οι μπορούμε να εφαρμοστούν για την αμοιβαιότητα αλλά και την ρήτρα προφύλαξη. Νομίζω ότι στη σημερινή συζήτηση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σημείο της μεσδιατάξεω για να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση πάνω και σε διαφορετικά ζητήματα. Όπως ε, εγώ δεν συμφωνώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία για οποιοδήποτε άλλο θέμα διεκδικήσεων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, μας απασχολεί εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει το ζήτημα της συμφωνίας με το βασίλειο του Μαρόκου ε, για πολλά ζητήματα όπως για τα βιολογικά προϊόντα στην ε, γεωργία θα μας αποσχολήσει όχι μόνο με, πάνω στο ζήτημα της ε, προέλευσης αλλά τώρα σε σχέση με την δράσεις του Μαρόκου σε σχέση με την ε, Σαχάρα. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το θέμα της μεσής διατάξης που θα μας απασχολεί εμείς. Θα πρέπει να περιοριστούμε σε κάποια ζητήματα μόνο. Το έπραξε σήμερα η Γενική Εύση Τρέιντ και Μάρε. Τώρα η Αλία από, από στενής ε, πλευράς δεν έχει καμία σχέση με το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει κάποια διαφορετική εταιρική συμφωνία Θεωρώ λοιπόν ότι στόχος της Επιτροπής μας είναι να ασχοληθεί με την αλληλευτική συμφωνία. Εκεί θα έχουμε πολλά να πούμε. Προς το παρόν δεν έχω να προσθέσω ρίποτε. Ευχαριστώ και μιλάμε. Ναι. Κατά άποψή μου δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ότι πρόκειται για μια καθαρά εμπορική συμφωνία. Εντάξει, προφανώς πρόκειται για μια εμπορική συμφωνία. Αλλά δεν πρόκειται ούτε για ενισχύσεις σε βοήθεια σε μια πιο φτωχή χώρα ή ούτε για μια ανθρωπιστική δράση. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας ε, καθαρής εμπορικής συμφωνία ε, από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου. Καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει αναγνωρίσει ότι η Δυτική Σαχάρα έχει την χάνει υπό την κυρία του Μαρόκου. Καμία χώρα. Και θα ήθελα λοιπόν οι πρώτοι που θα το πράξουν θα είμαστε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση διότι αυτό σημαίνει ότι προτάσουμε, μάλλον προτρέχουμε κάποιων αποφάσεων. Ξέρουμε ότι κάποιες, ε, κάποιες συμφέροντα υπάρχουν. Υπάρχει ενδιαφέρον της Ευρώπης ε, να αλλιεύει στις περιοχές αυτές, ε, προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους Ευρωπαίους εφοπλιστές που αλλιεύουν στην περιοχή. Εγώ είμαι υπέρ του να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή, αλλά πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το κλειδί της υποθέσεως και ισχύει για τα γεωργικά προϊόντα. Διότι και αυτό αφορά όλους, όχι μόνο την Επιτροπή Αλίας, την Επιτροπή ΑΦΕΤ την Επιτροπή Γεωργίας. Έχουμε μια θεμελιώδη αρχή ότι σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες με τις οποίες συνάπτουν συμφωνίες θα πρέπει να φέρουν το απο... να φέρουν το... τη σφραγίδα της σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαι πεπισμένος ότι στο Μαρόκο υπάρχουν και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και ο σεβασμός των ατομικών ελευθεριών. Αλλά στο Μαρόκο όλα αυτά. Αυτό δεν ισχύει για τη Δυτική Σαχάρα. Λοιπόν, αυτό είναι επιτακτικό για όλους μας σε ηθικό πρωτίστως επίπεδο και μετά σε εμπορικό. Λοιπόν, εάν στην περίπτωση αυτή η Δυτική Σαχάρα ο ε, συνομιλητή μας δεν σέβεται ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε τι ατομικές ελευθερίες. Υπενθυμίζω ότι το Κοινοβούλιο προ μερικών ημερών την περασμένη εβδομάδα ενέκρινε ένα, μια έκθεση που εισαγάγει και την χρήση των ε, φυσικών πόρων που βρίσκονται εκεί και που αφορά ε, ορυχεία αλλά και το ζήτημα των ε, ακτών. Πιστεύω λοιπόν ότι εμείς θα ασφάλουμε ως ε, Επιτροπή να ε, ξεπεράσουμε το ζήτημα με τρόπο απλό. Είμαι πεπισμένος ότι χρειάζεται από πλευρά Μαρόκου να υπάρξει η απόδειξη ότι τα πλεονεκτήματα φτάνουν στα χέρια των πληθυσμών. Αποδείξεις δεν έχουμε. Και εγώ σήμερα το πρωί ήμουν στην Επιτροπή Εξωτερικών που άκουσα τον πρόσωπο του μετόπου, του Πολυσάριο, θα πάω να ακούσω και τον πρέσβη του Μαρόκου. Στον πρόσωπο του Πολυσάριου δεν έκανα ερώτηση, αλλά θα θέσω ερωτήσει στον πρέσβη του Μαρόκου. Θα πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν πώ στο πλαίσιο αυτή τη συμφωνία μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε τι απαραίτητε προποθέσει για τον σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών των πληθυσμών. Εγώ δεν είμαι κατά τη συμφωνία, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε σεβόμενοι το δίκαιο σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχει πάρει και το Κοινοβούλιο μας, αλλά και σε ό,τι πρόκειται να προκύψει και από τις εμπορικές συμφωνίες ε, σε ύστερο στάδιο. Τώρα, το ζήτημα της αρχής. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σε αυτήν την Επιτροπή όσο και σε άλλες αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με τρόπο κατακαιρματισμένο. Ναι, άκουσα με προσοχή τον συνάδελφο, αλλά είναι δυνατόν να σκεφτούμε μια συμφωνία με τρία μέρη, όπου εμείς ε, ανανεώνουμε τις συμφωνίες, ε, αν κατάλαβα, αν καλά, ο Καντέκ λέει ότι κάνουμε συμφωνία, αλλά στο τραπέζι να βρίσκεται το Μαρόκο και η Δυτική Σαχάρα. Δεν είναι καινοτομία αυτό. Παρακάτω εδώ η Επιτροπή Εξωτερικών ακούει και το Μαρόκο και το μέτωπο του Πολυσάριου στην ίδια τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Ένα πράγμα είναι να ακούμε και το άλλο είναι να υπογράφουμε συμφωνίες. Μπορούμε να έρθουμε εδώ, να καλέσουμε όποιον θέλετε να μας ακούσει και να τον ακούσουμε, αλλά το να υπογράψουμε είναι άλλο πράγμα. Κύριε Σας ευχαριστώ. Λυπούμε που καθυστέρησα και αφήθηκα με καθυστέρηση. Ήμουνα στην Επιτροπή Εξωτερικών και άκουσα τον εκπρόσωπο της Δυτικής Σαχάρας ε, του Πολυσάριο και σε σχέση και με την ε, παρέμβαση του, του πρέσβη του Μαρόκου θα ακολουθήσει μετά. Δεν βρίσκω ότι ξεχωριστά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Δεν βρισκόμαστε σε ένα κενό υπενθυμίζω ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας και εκεί τονίζεται για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μια συνεκτική πολιτική ανάπτυξης πρέπει να ακολουθεί και να καλλιεργεί. Και ένας από τους πιο σημαντικούς κινητήρες ε, για το Μαρόκο είναι η πρόσβαση στους φυσικούς πόρους ε, του, της Δυτικής Σαχάρας. Αυτό έχει κέρια σημασία για το Μαρόκο και τα όσα συμβαίνουν εδώ παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Και αν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κινητοποιηθεί και δεν δράσει όπως κάνουν τα κράτη ΕΖΕΣ και όπως αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά οι όλα αυτά δηλαδή να αποκληθούν, αποκλειστούν από εμπορικές συμφωνίες όσα προέρχονται από κατεχόμενα εδάφη, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν κάνει κάτι τέτοιο θα νομιμοποιήσει αυτή τη στάση του Μαρόκου και δεν μπορούμε εμεί να συμφωνήσουμε φυσικά με κάτι τέτοιο να νομιμοποιηθεί αυτό. Αν είμαστε υπέρ λοιπόν τροποποιήσεων θα πρέπει να δεχθούμε το διεθνές δίκαιο και να το σεβαστούμε και δεν θα μπορούμε να σταυρώνουμε τα χέρια εδώ στην ε, δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να λέμε ότι τα θέματα αλληλεία ε, δεν ανήκουν στα ουσιοδέστερα θέματα διεθνούς δικαίου όσον αφορά το δίκαιο, τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα. Εδώ υπάρχει παράνομη κατοχή της Δυτικής Σαχάρας από τις, αρχές του, από τις δυνάμεις του Μαρόκου. Παρότι εδώ και πριν από 20 χρόνια ελήφθη αντίθετη απόφαση από τον ΟΗΕ. Εάν... Όπως είπε ο κ. Μάτος, ε, έχουμε μπλέξει δύο θέματα. Ένα πράγμα είναι το ζήτημα συμφωνία Μαρόκου με για το γεωργικό προϊόν και το άλλο είναι η συμφωνία Αλίας. Το, το ζήτημα της Γεωργίας ε, δεν το γνωρίζω καλά, αλλά βεστούσε αν ήταν επίση κάποια παρανομία τότε θα είχε γίνει καταγγελία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο συζητάμε εδώ, το κείμενο που συζητάμε εδώ δεν αναφέρει ότι είναι παράνομο, αλλά σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο θα πρέπει να γίνονται, δίνονται κάποιε αντισταθμίσει ε, κλπ. Ναι, ναι, μα έτσι έχει το πράγμα. Έτσι αναφέρει η γνωμοδότηση ε, νομική. Νομίζω λοιπόν ότι Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω είναι η συμφωνία Αλία. Τα άλλα δεν τα γνωρίζω πολύ καλά. Εν πάση όμω θα πρέπει να ξέρουμε πω σήμερα μα απασχολεί μια συμφωνία σύνδεση. Διότι δεν μιλάμε για την Αλία, δεν μιλάμε για την γνωμοδότηση που Μα αφορά. Σήμερα εκπρόσωποι της ε, Κομισιόν ή θα μας μιλήσουν για αυτή την ε, συμφωνία σύνδεσης ε, τώρα. Δώσω τον κύριο Ρωμέβα τον λόγο, αν θέλει να διατυπώσει κάποια ερωτήματα προς την Κομισιόν, αλλά παρακαλώ να επικεντρωθείτε στο ζήτημα των δύο μέτρων ελευθέρωση για τα γεωργικά προϊόντα και τα αντιευτικά προϊόντα. Δεν ξέρω αν θέλετε να θέσετε κάποια περαιτέρω ερώτηση προς την Κομισιόν. Ε, νομίζω ότι βρισκόμαστε εδώ σε ένα φαυλοκύκλο και από τον οποίο θα πρέπει να βγούμε. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα φαυλοκύκλο και πρέπει να διαρριχθεί αυτό ο φαύλο ε, κύκλο. Με κάποια επιχειρήματα θα, θα το δείξω αυτό για να απαντήσω στην ανησυχία τη Προέδρου. Αυτό που είναι νομική γνωμοδότηση και ο κύριο Καντέκα αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα νομίζω είναι σε σχέση με την ε, Συμφωνία Αλία. Συμφωνώ, δεν, είναι, δεν συσχετίζεται αυτό το θέμα με το σημερινό θέμα. Όμως ε, αυτό το οποίο λέει η γνωμοδότηση είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε αν το όφελος αυτών των πόρων έχει αντανάκλαση και έχει επιπτώσει, αλλά αν επίσης και είναι η επιθυμία των κατοίκων της Δυτικής Σαχάρας να λειτουργήσει αυτή η συμφωνία με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το δεύτερο τμήμα ξεχνάμε πολύ συχνά. Όχι μόνο ότι έχει επιπτώσεις, με θετικό τρόπο, αλλά να είναι και η βούληση και η επιθυμία των κατοίκων της Δυτικής Σαχάρας του Πολυσάριου. Και κανένας δεν διαρωτήθηκε γι' αυτό. Σημείο 2. Σε όσους ρωτήσαμε, είπανε σε σχέση με τους Σαχαράου ότι δεν έχουν πρόβλημα με τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εναντίον. Αλλά εδώ υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό. Δεν είναι εναντίον, αλλά οι διαπραγματευτές και οι υλοποιητέ αυτής της συμφωνίας, αυτό είναι το οποίο είναι το ουσιώδες. Δεν είναι κατά τη συμφωνία αλλά κατά του τρόπου που αυτή τη στιγμή είναι μια συμφωνία που ασκεί η κυβέρνηση του Μαρόκου εξουσία επιπόρων φυσικών που δεν τη ανήκει. Δεν τις ανήκουν, με συγχωρείτε. Αυτό είναι το θέμα. Είτε είναι τα φωσφατούχα, είτε είναι τα προϊόντα γεωργία είτε είναι τα, ε, τα προϊόντα αλεία. Δεν ανήκουν στο Μαρόκο. Γι' αυτό, γι αυτό ζητήσαμε την νομική γνωμοδότηση. Για να γνωρίζουμε αν υπό του σημερινού όρου η γνωμοδότηση για την αμοιβαία απελευθέρωση όσον αφορά γεωργικά και αλλιευτικά προϊόντα πραγματικά είναι νόμιμη και μπορεί να ε, θεωρείται ε, ότι έχει νομιμοποιηθεί. Και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις έχει υπογράψει συμφωνίες ε, απελευθέρωσης προϊόντων με τις ΙΠΑ για παράδειγμα το Μαρόκο, από την οποία συμφωνία αποκλείεται η επικράτεια της Δυτικής Σαχάρας, ρητά και κάθετα. Γι' αυτό λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση διατυπώνω την ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτησή μου. Να δούμε πώς εφαρμόζουμε τους κανόνες και κανονισμούς. Τελευταία και τέταρτη παρατήρηση. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να διαχωρίσουμε τα θέματα πράγματι. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε ως Επιτροπή Αλίας να, να ξεχνάμε ότι πέρα από το ότι είμαστε ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Αλίας, είμαστε ευρωβουλευτές μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναμένεται λοιπόν συνεκτικότητα στις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Όταν κάνουμε λόγο για αλία, δικαιώματα του ανθρώπου, είτε πρόκειται για μεταφορέ είτε άλλα θέματα, πρέπει τα δικαιώματα του ανθρώπου και το δίκαιο να λαμβάνονται υπόψη. Να είμαστε υπεύθυνοι και να είμαστε συνεκτικοί για αυτά τα θέματα. Δεν απαντήθηκαν τα ερωτήματα που έκανα και πρέπει να απαντηθούν. Γι' αυτό αναμένουμε την νομική γνωμοδότηση που ζήτησε ο κύριο Ζωζέ Μποβέ από την, ε, τις νομικές υπηρεσίες ε, και να ε, υποβληθεί αυτή και έτσι ελπίζω ότι θα εμβαθύνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Και μια τελευταία παρατήρηση. Όταν λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εξετάζεται ότι τα προϊόντα αυτά υπό το πρίσμα της αλληλείας είναι αλλιεύματα τα οποία έχουν αλλιευθεί από ε, μαροκινά πλοία ή από ευρωπαϊκά πλοία να μας το πούν αυτό ρητά και κάθετα. Αναφέρθηκε εδώ ένα θέμα και από τον κύριο Κάντα εδώ έχω την εντύπωση εγώ και εμένα και επιμένω ότι ανησυχεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση από το Μαρόκο. Έχει σχετικό μικρό βάρος το Μαρόκο και μεγαλύτερο βάρος η Ευρωπαϊκή Ένωση και την αφορά περισσότερο αυτό. Δεύτερον, αληθεύει ότι η σημαία ή τουλάχιστον η σημαία του πλοίου που αλλιεύει τα αλλιεύματα είναι σημαντικό. Αλλά επίση και από πού προέρχονται γεωγραφικά τα προϊόντα. Όταν αναλύουμε τη γεωγραφική προέλευση δεν αρκεί να καλύπτεται με τη σημαία του πλοίου, αλλά πού ακριβώ, σε ποια γεωγραφική ζώνη αλλιεύθηκαν αυτά τα ψάρια. Διότι διαφορετικά παραβιάζουμε ουσιώδει ρήτρε του διεθνού δικαίου και δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Ευχαριστώ. Bueno, eh, Ωραία. Νομίζω πως ε, το νομικό ζήτημα δεν ε, διαφέρει από συμφωνία ή συμφωνία, είτε πρόκειται για απελευθέρωση είτε για ελευθερική συμφωνία. Εσείς μιλήσατε για νομικές εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις κλπ. Τι θα πρέπει να προσδοκάμε από όλα αυτά. Α, το, το, ρωτάρε την Κομισιόν. δεν, δεν ξέρετε ότι υπάρχει κάποια γνωμοδότηση νομική, γιατί έτσι καταλάβαμε αυτά που είπατε. Όχι, εγώ αναφέρουμε σε αυτό που έκανε η Επιτροπή Ίντα, το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, απευθύνομαι προς την Κομισιόν νομικές γνωμοδοτήσεις ε, συντάσσει η Κομισιόν εάν καταρτίζει κάποιες ε, νομικές ε, γνωμοδοτήσεις. Μπορείτε να μου απαντήσετε παρακαλώ, είναι τα ή Γενική Διευθυνσή Μάρε, εάν υπάρχει κάποια νομική γνωμοδότηση στα σκαριά που φαίνεται κάτι σχετικό ο κύριος Δρομέδα ενώ εμείς οι υπόλοιποι αγνοούμε και που αφορά αυτήν την συμφωνία που μας απασχολεί για τη συμφωνία αυτή. Υπάρχει κάποια νομική γνωμοδότηση α, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ερώτηση, περιμένω απάντηση. Δυστυχώς θα σας απογοητεύσω, αλλά δεν ε, ετοιμάζεται αυτή η νομική γνωμοδότηση, αλλά δεν έχω στοιχεία. Βεβαίως ζητήθηκε στην Επιτροπή Ίντα και νομίζω ότι η Επιτροπή ΙΝΤΑ θα λάβει μια απάντηση σε αυτήν την ερώτηση στο αίτημα αυτό. Ε, δεν είμαι σε θέση να σας πω τώρα. Υπάρχει, ή αλλιώς να κλείσουμε τη συζήτηση αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ε, γνωμοδότηση νομική για την εμπορική συμφωνία και αναφέρομαι στα όσα είπε ο συνάδελφος. Υπενθυμίζω ότι μία νομική γνωμοδότηση ζητήθηκε εν ευθέτω χρόνο σχετικά με την αλλιευτική ε, συμφωνία και ότι η συμφωνία αυτή αφενός ε, δεν προσδιόριζε το πρόβλημα και δεν προκαταλάμβανε το πρόβλημα αυτό. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η συμφωνία, και θα πρέπει να το υπενθυμίσουμε, είναι οι σχέσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Μαρόκο. Ο εταίρος μας είναι το Μαρόκο. Με αυτόν διαπραγματευόμαστε και αυτό το θέμα το οποίο είναι κατανοητό, το οποίο το έχουμε εντάξει στον προβληματισμό μας αποτελεί ε, το αντικείμενο μιας ε, σειράς ε, επαφών για να έχουμε συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έχουμε όντως ζητήσει από τις αρχές του Μαρόκου μια σειρά ε, πληροφοριών, στοιχείων για τις διάφορες χρήσεις των μέσων, του μέσου του χρηματοοικονομικού που συνοδεύει αυτήν την συμφωνία και περιμένουμε, εξετάζουμε το θέμα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Κομισιό ενδελεχώς θα εξετάσει το θέμα προτού αρχίσει ε, τις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του πρωτοκόλου αυτού. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να τονίσω είναι οι κανόνες προέλευσης για τα αλλιευτικά προϊόντα είναι η σημαία του αλλιευτικού πλοίου. Αν πρέπει να βρούμε ένα άλλο κριτήριο, ε, υπάρχει ισορροπία γεωπολιτική όλης της πολιτικής μας. Αν ε, παίρναμε άλλα στοιχεία για να δώσουμε, για να προσδιορίσουμε την προέλευση ενός προϊόντος, ε, θα ήταν περίπλοκο. Για να επιλύσουμε λοιπόν ένα πρόβλημα σημαντικό ε, στα μάτια όλων μας, θα μπορούσαμε έτσι ε, να διακινδυνεύσουμε μια πολιτική που αντιπροσωπεύει πάνω από 55 δισεκατομμύρια κύκλο εργασιών. Σχετικά με τους κανόνες προέλευσης και την αναγκαιότητα μια συζήτησης, θα έχουμε ένα ραντεβού για την επόμενη συζήτηση, την προσεχώς, που θα λάβει η χώρα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης κοινή αλλιευτικής πολιτικής και τη μεταρρύθμιση του σκέλους αγορά. Επιτρέψατε μου να κάνω λίγη διαφήμιση για αυτό το στοιχείο της μεταρρύθμισης, εφόσον θα λάβει η χώρα σε μερικούς μήνες βάσει συγκεκριμένων προτάσεων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα να το κάνουμε νωρίτερα διότι το ζήτημα των ε, κανόνων προέλευσης είναι κάτι το οποίο θα προτιμούσα να συζητήσω με εσά και την Γενική Διεύθυνση Trade. Διότι εγώ συμφωνώ με εσά, αλλά με την Trade δεν συμφωνώ σχεδόν σε τίποτα. Ευαισθητός πρόκειται για μια νομική γνωμοδότηση που ζήτησε η Επιτροπή Ίντα για τη Συμφωνία Σύνδεσης. Ελπίζουμε λοιπόν, ε, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μας ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε, να δούμε τι θα κάνει η Επιτροπή Ίντα, πότε θα ψηφίσει κλπ. Εσείς προβλέπατε να συζητήσετε την έκθεση σας τον Ιανουάριο και η ψήφιση τον Μάρτιο και στην Ίντα. Επίσης ε, στα μέσα Μαΐου θα ψηφιστεί. Δώστε τον λόγο στον κύριο Καντέκ ε, τώρα αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με την ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν, ό,τι και να λέει η νομική γνωμοδότηση, εμείς το έργο μας θα πρέπει να το προχωρήσουμε. Κύριε Καντέκ, ε, παρακαλώ και να ολοκληρώσουμε. Δεν θα μακρηγορήσω, δεν ξέρω αν ε, δεν εκφράστηκα σωστά ή δεν έγινα απόλυτα κατανοητός. Δεν νομίζω πως είπα πως χρειάζεται να διαπραγματεύσουμε, να διαπραγματευτούμε τρεις γύρω από το τραπέζι. Απλά είπα θα πρέπει να επαληθεύσουμε ότι οι κλαδικές ενισχύσεις ε, καλύπτουν όλη την επικράτεια συμπεριλαμβανομένες και τις ε, περιοχές που κατοικούν οι Σαράουι. Όλοι λοιπόν θα χρειάζεται να ε, υποφεληθούν από αυτές τις συμβουλές. Είπα από την Ταγκέρη στο Μαλιμπού. Δεν είπα ότι πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση σε επίπεδο τριών. Είπε ότι είναι μια συμφωνία ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό. Περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 14, που αφορά την απόγραφηση αλίευση σε πραγματικό χρόνο για τη διαχείριση των αληθικών πόρων. Ο κύριος Νίκ Μπέιλ, ο κύριος Νέι του Ινστιτούτου των ε, του Θαλάσσιου Ινστιτούτο Επιστημών της Σκωτίας θα μας παρουσιάσουν μια έκθεση. Έχει, έχει διανυμηθεί ήδη το κείμενο, καλωσορίζω τους συγκεκριμένους και είναι το λόγο. Δεν ξέρω ποιος θέλει να λάβει το λόγο πρώτος, πάντως κάποιος από τους δυο σας αρχίσει. Uh, ευχαριστώ για αυτήν την εισαγωγή, κυρία ε, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που καλέσατε, ε, με καλέσατε και τον συνάδελφό μου Νίκ Μπέιλι ε, για το κρίσιμο σα σε πραγματικό χρόνο. Θα ήθελα να σας δώσω μια σύντομη εισαγωγή ε, σχετικά με τον, ε, την διαχείριση, την χωρική ε, των αλλιευτικών χώρων, την ανάπτυξη στην Ευρώπη και να συζητήσουμε ένα πρόγραμμα που έχουμε στην Σκοτία και το πρόγραμμα για την αξιολόγηση, της κριτικές, τα, οφείλη, ωφέλη των όσων κάνουμε, την, τα απαιτήσει και να κλείσουμε την συζήτηση σχετικά με τα real-time closures of fisheries. Έχουμε δύο κατηγορίες και μέτρα που μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν έλεγχη εισρωών, έλεγχη εκροών ε, και να δούμε τι γίνεται ε, σχετικά με τις, τα όρια αλλιευμάτων και το ποσοστό σχετικά με το φύλλο. Έχουμε τα εργαλεία έλεγχο χώρων, ε, output controls ε, εκροών, έχουμε τους περιορισμό αλίευσης, ε, ποσοστώσεις, μέγεθος εκφόρτωσης, ελάχιστο μέγιστο, σύνθεση αλιεύματος και το ποσοστό φύλου. Σχετικά με την με την ειδική ε, διαχείριση των χώρων αλίευσης. Έχουμε ε, διάφορες ε, περιορισμούς, περιορισμούς σχετικά με τα εργαλεία, τα αλλιευτικά που χρησιμοποιούνται και αυτό μπορεί να κατανοηθεί από τον κλάδο. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση μερικά χρόνια τα νησιά Φαρόε χρησιμοποίησαν ένα ειδικό σύστημα διαχείρισης χώρου και μπορείτε εδώ να δείτε ότι οι χώροι γύρω από τα νησιά έχουν ε, ουδέτερες, ουδέτερους χώρους, χώρους όπου είναι κλειστοί στην αλληλεία εδώ έχουμε ένα παράδειγμα από την ε, Δυτική Σκοτία ε, και για να ε, παρά για να έχουμε το, για να, την, το windsock, κλειστές περιοχές, μεγάλες περιοχές με ένα χώρο όπου ελέγχουμε τα εργαλεία αλίευσης και βλέπουμε ποιοι είναι οι περιορισμοί. Αυτό περιλαμβάνεται στην ε, διαδικασία την, ε, και στην νομοθεσία την ευρωπαϊκή. Βεβαίως ο κλάδος ε, δεν χαίρεται σχετικά με τα, τα μέτρα που υπάρχουν επιτόπου. Ένα πιο ευέλικτο σύστημα εξετάστηκε αλλά ε, δεν εφαρμόστηκε ε, διότι η ε, μεταποίηση, η επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο ήταν μια πρόκληση σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης. Πρόσφατα αυτές οι ανησυχίες διαλύθηκαν και έχουμε σε διάφορα μέρη του κόσμου μια εφαρμογή αυτού ε, του συστήματος. Ε, η Ισλανδία άρχισε να χρησιμοποιεί τα real-time closures ε, στη δεκαετία του 90 με επιθεωρήσεις αλλιευμάτων από δημόσιους κρατικούς παρατηρητές σχετικά με τις απορρίψεις. Αυτό είχαμε 120 απαγορεύσεις για τα τελευταία χρόνια. Επίσης, τα real-time closures χρησιμοποιούνται από την Νορβηγία και βασίζονται σε δείγματα που έχουν συλλεγεί και από περιοχές που περιλαμβάνουν ε, υπερβολικό ποσοστό γόνων. Ε, τα λεπτομέρειε του προγράμματος περιλήφθηκαν σε διμερείς διαπραγματεύσεις υποστηρίζεται το σύστημα αυτό από τις νορβηγικές αρχές ούτω ώστε να μπορούν να ανασύσταθούν τα αποθέματα γάδου στην περιοχή. Δεν υπάρχουν συντονισμένες προσπάθειες στην Ευρώπη αλλού, παρόλο που μεμονωμένα κράτη έχουν υιοθετήσει δικά τους προγράμματα. Ε, κυρίως για το γάδο ε, ούτως ώστε να ανασυσταθούν και στη Βόρεια Θάλασσα ε, τα αποθέματα. Η Αγγλική ε, Διοίκηση, η Γαλλική επίσης έχουν ασχοληθεί και στην, για την περιοχή Κάτεγκάτ. Επίσης έχουν καταβλεθεί προσπάθειες. Στην Σκοτία έχουν, το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί το 2008 εισήχθη για να περιορίσουμε στο χώρο, για περιορισμούς το 2009 επεκτάθηκε ούτω ώστε να μειώσουμε κατά 25% την θνησιμότητα. Αυτό είναι η χρονική περίοδος. Στο 2007 για να μειώσουμε την θνησιμότητα σχετικά με τον γάδο του 2005. Έχουμε κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία. Στο Συμβούλιο υπήρξε μια συμφωνία τα κράτη-μέλη ε, να επεκτείνουν τέτοια προγράμματα, να τα διευρύνουν. Η ε, μόνιμη επιτροπή, η μόνιμη ομάδα συστάθηκε το 2008 και περιλαμβάνει εκπροσώπους του αλληλευτικού κλάδου, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιστήμονες. 2008 για την ε, προστασία του γόνου και του γάδου Βάσει των ε, παρατηρήσεων και τον Νοέμβριο 2008 η STCF θεώρησε ότι το πρόγραμμα είναι μια προσπάθεια θετική, αλλά ότι χρειαζόταν να διευρυνθεί για να έχει αντίκτυπο θετικό. 2009 οι υπολογισμοί έδειξαν 10 ε, φορές ε, περισσότερες απαγορεύσεις και για την μείωση της θνησιμότητας και ένα σύστημα υπολογισμού ε, εξετάστηκε. 2009 ε, 144 απαγορεύσεις, το 2010 συνεχίστηκε το πρόγραμμα αυτό. Εδώ μερικές λεπτομέρειες του προγράμματος υπάρχουν ε, μέσα ε, για το κλείσιμο αυτό σε πραγματικό χρόνο, για την απαγόρευση. Έχουμε ορισμένες ε, στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν τον υπολογισμό, τον υπολογισμό του μέσου αλλιεύματος. Γίνονται επιθεωρήσεις στην ανοιχτή θάλασσα. Επίσης, ορισμένες δηλώσεις από τους ίδιους τους keepers, τους καπετάνιους. Ε, πώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Από το 2008 ε, καλύψαμε μια ε, περιοχή 56 τετραγωνικών ναυτικών μιλίων και βλέπουμε ότι πέρσι υπήρξε τέσσερις φορές μεγαλύτερη απαγόρευση όπου υπάρχει μια απαγόρευση δίπλα σε έναν αγωγό ε, πρέπει ε, να προσαρμοστεί καταλήλως. Έχουμε ε, διάρκεια 21 ημερών αυτόματη επανέναρξη. Λαμβάνονται οι αποφάσεις από το, τη μόνιμη επιτροπή, την οποία ανέφερα, όταν αρχίζει μια απαγόρευση, η τοποθεσία αυτή ανακοινώνεται στα πλοία, ούτως ώστε να ξέρουν ε, ποιο, ε, ποια περιοχή θα κλείσει στην αλία. Ε, έχουμε ιστότοπο, επίσης που περιλαμβάνει χάρτη με όλες τα, τους χώρους και τα σημεία της περιοχής απαγόρευσης, ούτως ώστε να δει κανείς το Μάιο βλέπετε που ε, εδώ ε, ποιες περιοχές ε, έχουν απαγόρευση. Έχουμε εδώ τετράγωνα μαύρα και κίτρινα, μπορείτε να δείτε. Βλέπετε περιοχές όπου δεν μπορεί να υπάρξει μια άλλη απαγόρευση, ούτως ώστε να μην υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση ενός συγκεκριμένου κλάδου. Βλέπετε επίσης κόκκινες γραμμές ε, που περιχαρακώνουν τις ε, περιοχές ε, στην δυτικά της Σκοτίας, ούτως ώστε να έχουμε καλή κάλυψη και να δούμε ποιος αριθμός απαγορεύσεων θα υπάρξει σε αυτές τις περιοχές σχετικά με την παρακολούθηση για να δούμε την συμμόρφωση Η συμμόρφωση αυτή παρακολουθείται, επιτηρείται από στοιχεία VMS ε, και υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχουν ε, ποινές, ε, κυρώσεις, μια κύρωση πέντε ημερών γενικά για παραβίαση το 2009. Επιστολές απεστάλησαν σε πλειοκτήτες 21 πλοίων. Υπήρξε κύρωση μία φορά σε 7 πλοία και ένα πλοίο υπέστη κύρωση δύο φορές. Εδώ έχουμε ένα χάρτη της τοποθεσίας των, των περιοχών απαγόρευσης το 2009. Βλέπουμε ότι στην, πώς ακολουθούν την υφαλοκρηπίδα και βλέπουμε ότι πώς ακολουθούν τα κόκκινα τετράγωνα είναι απαγορεύσεις και κίτρινο και πράσινο ε, βλέπουμε εδώ τι έχουμε παρατηρήσει σχετικά με τα πλοία 2010, η ίδια εικόνα που δείχνει την τοποθεσία των απαγορεύσεων, καφέ μικρότερης, μικρότερου μεγέθους και, ε, ε, και πράσινο μεγαλύτερου μεγέθους. Μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των απαγορεύσεων σε πραγματικό χρόνο είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι δύσκολο να, περιλα... να, να προβλέψει κανείς. Πρώτα απ' όλα ε, πρέπει να εντοπίσουμε ε, τις, ε, τους χώρους απαγόρευσης, τις περιοχές απαγόρευσης. Σας το έδειξε αυτό. Έχουμε στη Βόρεια Θάλασσα τα στοιχεία που δείχνουν πληθώρα γάδων και στα ε, δυτικά ε, της Νορβηγίας και πλησίων των νησιών Σέτλαντ. Έχουμε λοιπόν κάποια εμπιστοσύνη ότι αποδίδουν τα μέτρα αυτά. Δεύτερον, είναι σωστή η έκταση ε, των περιοχών απαγόρευσης. Εδώ έχουμε την αποθήκευση διαφόρων ε, στοιχείων σχετικά με το γάδο και βλέπουμε τις κινήσεις διαχρονικά και βλέπουμε τι ποσοστό γάδων έχουν ε, παραμείνει ε, στο πλησίον του σημείου. Έχουμε εδώ τις περιοχές, περιοχές απαγόρευσης ότι σε 21 μέρες ε, λιγότερο από μισή γάτη παρέμειναν στην σε αυτές. Εδώ με κίτρινη γραμμή βλέπουμε ότι περίπου 75% παρέμειναν ε, των γάδων στην περιοχή ε, στην ίδια περίοδο. Επίσης το θέμα που απασχολεί είναι η έκταση των περιοχών απαγόρευσης. Μήπως αυτές μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά ε, των αλλιευτικών πλοίων. Τα προγράμματα αυτά εδώ 7 μέρες ε, πριν και κατά τη διάρκεια ε, της έρευνας και της απαγόρευσης βλέπουμε υπάρχει πολλή αλίευση στην περιοχή που θα, όπου θα απαγορευτεί η αλία και μετά έχουμε ε, μετακίνηση ανατολικά και δυτικά. Δεν ξέρουμε αν τα πλοία αλλιεύουν στα όρια της περιοχής απαγόρευσης. Βλέπουμε ότι μετακινούνται σε άλλες περιοχές. 9 φορές στις 10. Τέλος και το σημαντικότερο υπάρχει επιτυχία στην μείωση της θνησιμότητας των γάδων. Αυτό το, το στοιχείο μας δείχνει ε, τους διαθέσιμους γάδους για τον στόλο ε, της Σκοτίας. Αυτή είναι μια εκτίμηση της συνολικής θνησιμότητας γάδων. Έχουμε τις απορρίψεις πάνω το γκρι είναι από το 2008 η αλίευση και έχουμε 25% μείωση στη θνησιμότητα. Εδώ έχουμε τις εκφορτώσεις που αναφέρθηκαν από τον στόλο, τον σκοτικό. Οι απορρίψεις βλέπουμε ότι τα αλιεύματα και οι εκφορτώσεις οδήγησαν ε, στη μείωση 25% της θνησιμότητας που ήταν ο στόχος μας. Πρόκειται για ένα ε, αντιδραστικό πρόγραμμα. Ε, τα στοιχεία βασίζονται σε αλλιεύματα που ήδη υπάρχουν και όχι σε ε, προβλέψεις. Βασίζονται σε στοιχεία VMS, βασίζονται στα, στις, ε, στους κανονισμούς VMS, ε, αλλά υπάρχουν μερικά πλοία τα οποία είναι πολύ μικρά και δεν, έχουν, δεν είναι εξοπλισμένα με VMS. Νομίζω ότι θα πρέπει τα μελλοντικά στοιχεία να μας βοηθήσουν σε καλύτερη εκτίμηση και τελικά κυρώσεις ε, για παραβίαση αυτών των real-time closures ε, μπορούν να υπάρξουν για σκοτικά πλοία, η δραστηριότητα από μη σκοτικά πλοία είναι άγνωστη ποσότητα. Έχουμε εκφορτώσεις που δεν ξέρουμε από πού ε, προέρχονται. Υπάρχει βεβαίως μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Δείξαμε ότι πρέπει να έχουμε, για να βελτιώσουμε τις τεχνικές απαιτήσεις, να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο, ε, να έχουμε καλύτερη προσέγγιση της διαχείρισης, οι κυβερνήσεις και οι αρχές. Ε, θα πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα και να έχουμε επίσης τεχνικές διαδικασίες και επεξεργασίες. Κλείνοντας, θα μπορούμε να δούμε, να υποθέσουμε σε ποιες περιοχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα προγράμματα ε, real-time ε, closures ε, για την αναπαραγωγή βορειοδυτικά στη σκοτίας για να προστατεύσουμε την αναπαραγωγή και τους γόνους. Επίσης, έχουμε μια προστασία ε, για την Πεσκανδρίτσα και εδώ έχουμε επίσης, εδώ που περιοχές αναπαραγωγής, εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Βεβαίως, η προστασία, ε, πρέπει να έχουμε στο θαλάσσιο περιβάλλον και προστασία ε, για διάφορες μεταναστεύσεις ορισμένων θαλασσίων θηλαστικών, ας πούμε, ε, η χρήση σε ένα ε, περιβάλλον, σε ένα πλαίσιο που υπάρχουν πάρα πολλά είδη ε, και απορρίψεις θα μπορούσαν να κλειστούν ορισμένε περιοχές, να υπάρξει απαγόρευση και για να προστατεύσουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των αλλιευτικών προϊόντων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτό όπως και στον κόλπο του ε, Μεξικού. Επίσης, ε, με παρακολούθηση καθημερινή, χρησιμοποιώντας δορυφορικά στοιχεία, για να, όπως έγινε εκεί στον κόλπο του Μεξικού για την πετρελαιοκυλίδα. Ευχαριστώ πολύ. Gracias. Eh, Ευχαριστώ. Επιθυμεί κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο. Διαφορετικά εγώ έχω μερικές ερωτήσεις να σας θέσω. Φυσικά είμαστε λιγοστοί στην αίθουσα, αλλά αυτό οφείλεται στη συζήτηση που διεξάγει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Κύριε Κούν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Είδαμε πως εργάζεστε πραγματικά με ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο για την προστασία των αποθεμάτων και πως η, ε, ε, η επαγγελματική αλληλεία αντιμετωπίζει το ζήτημα με ιδιαίτερη σοβαρότητα όταν ε, ορίζεται περιοχές απαγόρευσης αυτό αποτελεί αναφίβολα ένα πλήγμα για τον κλάδο της αλίας. Εδώ για τον γάδο <clears throat> έχετε ένα τάκ, αλλά αυτό κοστίζει περισσότερο λόγω της ε, περιοχής απαγόρευσης. Οι περιοχές αλίας ε, ελέγχονται με τρόπο ιδιαίτερα αυστηρό, κάτι το οποίο μάλλον περιορίζεται, περιορίζονται με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο, κάτι το οποίο επιτρέπει έναν αποτελεσματικό έλεγχο. Και έτσι έχουμε ικανοποιητικέ δυνατότητες ε, αξιολόγησης της καταστάσεως και μπορούμε να ελέγχουμε κατά πόσον οι ποσοστώσεις ε, ε, χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό τρόπο κλπ. Τώρα πρέπει να δούμε κατά, κατά πόσο στη μεζόγειο, στην Θάλασσα ε, της κλπ. Υπάρχουν παρόμοια συστήματα παρακολούθησης. Ε, ε, μπορούμε να έχουμε λοιπόν μια γενικότερη άποψη που θα μπορούσε να αξιολογήσει τις ιδιαιτερότητες του αλλιεύματος, την πορεία της βιομάζας. Υπάρχουν λοιπόν μοντέλα τα οποία έχουν καταρτιστεί και που να καλύπτουν πολλές χρονιές που θα επιτρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με τον γόνο να υπολογίσουμε τον αριθμό των γόνων σε σχέση με τη βιομάζα, σε σχέση με τα συνολικά αλλιεύματα. Εδώ λοιπόν ερωτήματα που θα ήθελα να σας θέσω. Γι' αυτό λοιπόν έκανα ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και πιστεύω πως όλοι όσοι έχουν διαπραγματεύσει με το Μαρόκο έχασαν πραγματικά πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση. Ίσως να μην κατάλαβα καλά, να μην παρακολούθησα τη συζήτηση από το αρχείο στο τέλος, αλλά αυτές τις περιοχές απαγόρευση εφαρμόζονται σε, όλες τα, σε όλα τα σκάφη Α, και ε, αυτό μήπως αφορά μόνο τα σκάφη τα οποία θέτουν συστήματα παρακολούθησης σκαφών, VMS, Εδώ υπάρχει μια, ένας μύθος που λέει ότι τα μικρά σκάφη είναι πολύ καλά και τα μεγάλα όχι. Κάνουν, ε, τα μένουν πολύ καλά η δουλειά τους, τα άλλα κάθε άλλο παρά καλή, καλά εκτελούν το έργο τους. Ευχαριστώ. Να, να μου απαντήσετε και στις δύο ερωτήσεις. Uh, Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις σχετικά με την Πρόεδρο. Για την ώρα η ικανότητα ανιχνεύσεως που βρίσκονται να εντοπίσουμε ε, τα πλοία είναι δύσκολη. Μπορούμε να εντοπίσουμε τα μεγάλου μεγέθους πλοία. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι καλύτερα τα μικρά πλοία ε, και κακά τα μεγάλα, αλλά πρέπει να πούμε ότι ε, ε, οι μεγαλύτερες, ε, ο συνοστισμός, η πληθώρα των γάδων βρίσκονται στα άκρα της υφαλοκρηπίδας και γι' αυτό αλλιεύονται από τα μεγάλα πλοία. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε λοιπόν τη θνησιμότητα έχουμε κάποια αποτελεσματικότητα και υπάρχουν ορισμένες προβλέψεις για μέτρα για να παρατηρήσουμε, να παρακολουθήσουμε την απαγόρευση σε αυτές τις περιοχές. Καταρχήν, το rollout των VMS ε, νομίζω ότι είναι εποφελές για πάρα πολλές απόψεις της αλίας και όχι μόνο για τη θνησιμότητα των γάδων. Και νομίζω ότι έχουμε ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, σχετικά με την θνησιμότητα ορισμένων ειδών αλλά και με άλλα θέματα και με άλλους, άλλους τομείς σχετικά με την ε, διατήρηση. Σχετικά με την ερώτηση για την εφαρμοσιμότητα σε άλλες περιοχές και πάλι καταρχήν δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ε, σε άλλες ε, περιοχές αυτό το πρόγραμμα των real-time closures του, της απαγόρευσης σε πραγματικό χρόνο αυτό είναι μέρος ενός γενικότερου προγράμματος για την διατήρηση, αλλά κυρίως σε σχέση με το γάδο. Αν πάμε σε άλλες περιοχές που έχουν ε, διαφορετικούς στόχους και διαφορετικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα αυτό αναλόγως. Αλλά καταρχήν είναι εφικτή η χρησιμοποίηση του προγράμματος και αλλού και σε άλλους τομείς. Αναφέρθηκε ότι ε, πολλή εργασία περιλαμβάνεται σε αυτή τη δραστηριότητα, σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αυτό είναι αληθές και παρατηρούμε ότι ενώ αναπτύσσουμε το πρόγραμμα ε, θα πρέπει να ε, διευρυνθεί και να προσαρμοστεί, αν θέλετε, ο φόρτος εργασίας για αυτόν τον αυξήθηκε λόγω του μεγαλύτερου αριθμού ζωνών απαγόρευσης και το θέμα που παραμένει είναι η χρησιμότητα αυτών των real-time closures, των απαγορεύσεων σε πραγματικό χρόνο, αν είναι ένα είδος πανάκια, μπορεί να είναι βεβαίως ένα χρήσιμο αργαλείο, αλλά αν πρέπει ε, να έχετε στόχους ε, σημαντικούς για μείωση της θνησιμότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και άλλες μεθόδους. Είναι ένα στοιχείο ε, του εργαλειοκιβωτίου και όχι το μοναδικό στοιχείο, το μοναδικό εργαλείο. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Κούν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μια επερώτηση θα είχα. Μια και τώρα, για παράδειγμα, όσον αφορά το γάδο, ήταν υποχρεωτικό μέσω των περιοχών που έκλεισαν οι στόλοι να πάνε σε άλλες περιοχές να αλλιεύουν. Ποια συμπεράσματα έχετε συναγάγετε Ξέρετε ποια είναι τα κύρια, οι κύριες περιοχές αλλιευμάτων. Εμπειρικά ξέρουν που βρίσκεται το ψάρι, εκεί πάνε και εκεί πάνε και το πιάνουν το αλλιεύμα αυτό. Όταν υπεκφεύγουν και πάνε σε άλλες περιοχές, τότε αυτά τα νέα στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη για την συνολική βιομάζα και το ε, πρότυπο υπολογισμού. Και αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Κανονικά έχουμε μια κλίδα κανονικής κατανομής και μετά υπάρχουν παρεκκλήσεις από αυτό υπάρχουν κάποια στοιχεία, δίνονται κάποια στοιχεία για τη βιομάζα και τον υπολογισμό, για παράδειγμα, κάποιων αλλιευμάτων, των σπογκοδών για παράδειγμα. Yes, I'll, I'll try and answer Θα προσπαθήσω να απαντήσω οι πληροφορίε που χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση των αποθεμάτων και της βιομάζας και για την θνησιμότητα είναι προφορίες που λαμβάνουμε από τον κλάδο αλλά και από ερευνητικά σκάφη και από άλλα στοιχεία α, ανεξάρτητων αρχών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση από μια περιοχή σε άλλη, τι απαγορεύσει, αυτό εξαρτάται από τις πληροφορίε που έχουμε, αλλά συνεχώς υπάρχει, υπάρχουν κάποια ε, στοιχεία από ανεξάρτητες, ανεξάρτητες φορείς που μας βοηθούν στην γενικότερη προσέγγιση μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους δύο προσκεκλημένους για την ε, παρουσίαση του θέματος. Έτσι ολοκλώσαμε το σημείο 14 της και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, το υπαριθμό 15, που είναι τα πρακτικά της 17ης έκτακτης συνεδρίασης ε, της ε, ΕΚΑΤ ε, νομίζω ότι το εξετάσαμε χθε το ζήτημα αν δεν υπάρχει κάτι που να θέλει να προσθέσει να το τελευταίο σημείο της αφορά στην εντροσωπία της Επιτροπής Αλίας ε, στην Μαυριτανία. Όλοι οι βουλευτέ ε, θα θέλαν να μάθουν τι πράξαμε στη Μαυρτανία. Σας πω ότι η εξοπία στη Μαυρτανία, τη οποία ηγήθην εγώ, αποτελεί τον κύριο Καντέκ, του Λοβίν και Φερέιρα από την ε, Γκουε. Ε, καταρτήσαμε ένα πρόγραμμα με την διοίκηση της Μαυριτανίας και την τελευταία στιγμή ένα από τα σημαντικά σημεία που ήταν η επίσκεψη σε κάποιο λιμάνι που, ήταν το, που είναι το σημαντικότερο όλης ε, ε, της, όλης της ακτής της Βρετανίας ακυρώθηκε. Κάναμε όμως διάφορες επισκέψεις. Ε, είδαμε τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Αλίας Εν το πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ιδιαίτερα ευρύ και είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με πολλούς συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων του κλάδου ε, και του αεραστεχνικής αλίας ε, θα θέλαμε επίσης να μιλήσουμε και με τον κύριο Νάουα και όλο το προσωπικό της ε, πρεσβείας, ε, τους οποίους και ευχαριστήσαμε για την συνεργασία τους. Όπως γνωρίζετε, η Συμφωνία Λίας με τη Μαυριτανία είναι η σημαντικότερη που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες, ε, τόσο σε αφορά των αλλιεύματα όσο και την οικονομική πτυχή, το 50% του προϋπολογισμού που χορηγείται στην τομέα της ε, Αλίας ε, αφορά στην συμφωνία με τη Βρετανία. Επίσης πρόκειται για μια συμφωνία που περιλαμβάνει και αφορά τις ε, τους επιρροές ελευτικούς στολίσκους οκτώ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένα Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ελλάδας κλπ. Υπάρχουν λοιπόν πολλές Υπάρχουν πολλοί στόλοι των κρατών μελών και όχι ενός κράτους μέλους μόνο. Θέλω να υπογραμμίσω κάποια πράγματα για αυτή την επίσκεψη. Πρώτα απ' όλα, σαν ολοκλήρωση του ταξιδιού, το μεγάλο ενδιαφέρον που καταδείχθηκε από τις μαυριτανικές αρχές για την συνέχιση της Συμφωνίας Αλίας, τη συνέχεια της, που όπως γνωρίζετε πρέπει να την αναδιαπραγματευτούμε του χρόνου το 2011. Τα προβλήματα που υφίστανται, που είναι πολλά και ίσως πολλά που οφείλονται στο ότι η τελευταία διαπραγμάτευση δεν ήταν απόλυτα σωστή και ορθή. Πολλά όμως από αυτά επιλύονται, ιδιαίτερα όσον αφορά τα αλλιεύματα και την επιβολή κυρώσεων που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαμε με αυτή τη συμφωνία. Και μετά από την ε, μεικτή επιτροπή που έγινε το Φεβρουάριο πέρσι φαίνεται ότι υπήρξε θετική αντίδραση από πλευρά ε, των μαυριτανικών αρχών. Και αυτό το θέμα που μα ε, μας ανησυχούσε ιδιαίτερα, ανησυχούσε Στου στόλους βελτιώθηκε. Όσον αφορά την οικονομική αντιστάθμιση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Μαυριτανία, 30% είναι <clears throat> όσον αφορά τα έσοδα από πλευρά τη δημοσιονομική ε, των εσόδων, 30% είναι ε, αντιστάθμιση οικονομική τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ τη Μαυριτανία. Και από αυτό μπορείτε να συναγάγετε τη σημασία που έχει για του Μαυριτανού υπό την οικονομική πλευρά η Συμφωνία Αλία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και το συμφέρον που είχαν οι αρχές της Μαυριτανίας να έχουμε μία επαφή με τον Υπουργό Οικονομικών που πραγματικά προσπάθησε να μας δώσει όλες τις διασφαλίσεις που μπορούσε, που ήταν δυνατόν, για την χρηματοοικονομική αντιστάθμευση, κυρίως εκείνη που στόχευε στην τομεακή ανάπτυξη για την ανάπτυξη της Αλίας και του στόλου στη Μαυριτανία. Η Υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να πω, μια, ένα θέμα για τη χρήση αυτών των κονδυλίων που πρέπει να γίνει σωστά. Μια άλλη πτυχή που εξετάσαμε με τις αρχές της Μαυριτανίας, αλλά όχι με μεγάλη επιτυχία, ήταν το θέμα του ότι άλλες, άλλοι στόλοι τρίτων χωρών αλλιεύουν στην ίδια περιοχή. Όπως γνωρίζετε, σαν συνέπεια του διεθνούς δικαίου, οι στόλοι που αλλιεύουν σε, ένα, σε μια αλλιευτική περιοχή οικονομικής αποκλειστικής ζώνης μιας χώρας καταρχήν πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τα πλεονάσματα, μόνο τα πλεονάσματα σε σχέση με την ε, χρήση του στόλου ή της αλλιείας μιας συγκεκριμένης χώρας, σε αυτή την περίπτωση της Μαυριτανίας. Έπρεπε λοιπόν να δούμε ότι αλλιεύουν άλλοι στόλοι εκεί, να δούμε ποια είναι τα πλεονάσματα και πώς θα κατανεμηθούν τα πλεονάσματα. Αυτό ήταν ένα ταμπού ως θέμα Κανένας δεν το έφυγε. Και παρότι έχουν, έχει, είχε τεθεί επανειλημμένα, δεν υπήρχε αντίδραση και απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, στο ταξίδι στην αποστολή είδαμε σε σχέση με κάποιους τομείς, όχι τον ισπανικό τομέα, αλλά τομείς άλλων κρατών μελών που ε, δεν αναφέρω. Θέλω να πω ότι ετοιμάζεται μια συμφωνία από πλευρά τους με την Κίνα. Η Κίνα έχει συμφέρον, έχει πολλά συμφέροντα εκεί παρότι το μεγαλύτερο μέρος των στόλων της Κίνας ε, υπό σημαία της Μαυριτανίας ε, αλλιεύει. Θέλουν όμως οι Κινέζοι να κάνουν μια νέα συμφωνία με τη Μαυριτανία σχετικά. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι σημαντικό θέμα να το λάβουμε υπόψη με τις, για τις διαπραγματεύσεις. Και παρότι σας λέω, παρότι δεν συναγάγαμε μεγάλα συμπεράσματα και δεν, βρήκαμε, δεν μας δώσανε μεγάλα στοιχεία για αυτά. Ε, υπάρχει αυτή η αυτό το στοιχείο της αλίευσης από άλλους τόλους ε, της Κίνας, ε, των Ρώσων, της Ουκρανίας. Φαίνεται ότι οι Κινέζοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Άλλα προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν και υπογραμμίζω αυτή την πτυχή είναι το πρόβλημα των επενδύσεων. Ζήτησαν περισσότερε επενδύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι Μαυριτανοί. Παραπονέθηκαν, για παράδειγμα, ότι τα μεγάλα σκάφη με γρήπου, πελαγικά ε, σκάφη, πάνε και ξεφορτώνουν στην Λασπάλμα των Καναρίων νήσων απέναντι από τη Μαυριτανία. Το λέω αυτό για να δείτε γεωγραφικά τι συμβαίνει. Πάνε, αντί να πάνε στο λιμάνι του Νουαντίμπου, πάνε στο Λασπάλμα των Καναρίων νήσων. Αυτό συναρτάται με τις υποδομές που δεν έχει η Μαυριτανία. Οι επενδύσεις ε, θα πρέπει να συνδέονται φυσικά με την ανάπτυξη των υποδομών που αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναπτυχθεί. Το πιο σημαντικό λιμάνι εκεί είναι το λιμάνι Νουαδιμπού που ε, έχει ακριβώς και την, ε, αυτή, την, ε, την πλευρά του Μαρόκου από την άλλη πλευρά. Είναι ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξή του που χρηματοδοτείται από την Ισπανία. Λένε ότι σε δύο χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Εδώ 20 χρόνια εγώ το, τα παρακολουθώ τα πράγματα και έχω αμφιβολίες αν μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Και υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα για το λιμάνι του Νουαδιμπού. Η βήθηση, η καταβήθηση είναι σκάφη τα οποία έχουν βυθιστεί, ε, δηλαδή θα λέγαμε ναυάγια στο αγκυροβόλιο του λιμανιού. Πολλά ναυάγια και έτσι η πρόσβαση στο λιμάνι είναι σχεδόν ανέφικτη, είναι επικίνδυνη. Και έτσι λοιπόν οι, ε, όλες οι εργασίες γίνονται στην έξοδο, στην είσοδο του λιμένα για να αποκτήσει τη σημασία που πρέπει να έχει και όλοι επιθυμούμε να έχει αυτό το λιμάνι πρέπει οι εκφορτώσεις που γίνονται στις, και να γίνονται οι εκφορτώσεις αντί στις Λασπάλμα στον Ουαδιμπού πράγμα που θα είχε πρόσθετη αξία για τους Μαυριτανούς, είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθούν αυτά τα προγράμματα και αυτά τα σχέδια, να αποσυρθούν, να ανελκυστούν τα ναυάγια, να καθαριστεί το λιμάνι, να αποκτήσει υποδομές. Αυτό επιμείναμε και είπαμε στις αρχές της Μαυριτανίας. Υπάρχει ένας τομέας, ε, ένα μέρος του τομέα για την εκφόρτωση ε, στην Λασπάλμας που εξετάζει τη δυνατότητα επενδύσεων επενδύσεων ε, στον Και αυτοί όμως απέτυσαν, αυτό ο τομέα απέτυσε να ολοκληρωθεί το έργο του Λιμένα το δυνατόν πιο νωρί ε, και για να μπορέσουν τέτοια προγράμματα να λειτουργήσουν. Αυτό το θέμα των υποδομών είναι ένα θέμα θεμελιώδου σημασία. Κρίμα είναι που όλα αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Πόσο μάλλον επιπλέον τα χρήματα για την τομεακή ανάπτυξη δεν χρησιμοποιούνται τα κονδύλια αυτά πλήρως ε, όσον αφορά τους Μαυριτανούς. Ελπίζουμε όμως ότι σε μια προθεσμία δύο ή τριών ετών τα προβλήματα κυρίως στο λιμάνι του Νουαντιμπού θα επιληθούν και θα είναι πιο εύκολο για τα κοινοτικά σκάφη να μπορούν να εκφορτώνουν εκεί και να γίνουν και οι αναγκαίες επενδύσεις. Ένα άλλο θέμα είναι του ελέγχου <clears throat> μέσω της υπηρεσίας ε, για την παρακολούθηση αλίας. Ξέρετε ότι στην τελευταία συμφωνία αλίας που υπεγράφει με τη Μαυριτανία η Ευρωπαϊκή Ένωση επέμεινε όπως επιμένουν, επιμένουμε σε όλες τις συμφωνίες με τρίτες χώρες για τη σημασία που έχει ο έλεγχος ε, όσον αφορά τα αλλιεύματα την υπηρεσία αλίας. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, όπως για παράδειγμα οι, τα δικά μας σκάφη κινούνται και αλλιεύουν ε, σε συγκεκριμένες ζώνες. Ο έλεγχος σε τρίτες χώρες πρέπει να γίνεται από τους ε, επιτηρητές, τους επόπτες. Υπήρξε ευρεία συζήτηση που διεξήχθη έχει, είχε αντικατασταθεί σε σχέση με τον έλεγχο αλλά έχει τεθεί και πάλι αυτό. Παρότι η Μαυριτανία έχει υπογράψει ένα πρωτόκολλο με την υπηρεσία αυτή. Λένε όμως οι Μαυριτανοί ότι δεν είναι αξιόπιστη 100% λέει η υπηρεσία αυτή. Κανένα σύστημα δεν είναι 100% ε, αξιόπιστο βέβαια. Λένε ότι υπάρχουν άλλα εναλλακτικά συστήματα όπως ο έλεγχος με το ραντάρ, η καταχώρηση και η αναφορά στις ε, υπηρεσίες Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα το οποίο επισημάνθηκε στις αρχές των Μαυριτανών είναι ότι μπορούν να λένε ότι ε, δεν είναι το καλύτερο σύστημα ελέγχων αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι όμως απαράδεκτο είναι να έχουμε άλλα εναλλακτικά συστήματα τα οποία δεν δίνουν νομική ασφάλεια σε κανέναν, δεν δημιουργούν νομική αξιοπιστία. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο πάλι θα πρέπει να το δούμε και επανήλθαμε σε αυτό είπαμε σε σχέση με τους Μαυριτανούς ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα αυτό των ελέγχων είναι θέμα αρχής και γι' αυτό θα πρέπει στο μέλλον να δουν πώς θα μπορέσει να γίνει και να λειτουργήσει όλο αυτό το πλέγμα, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα αυτό θα μπορεί να λειτουργήσει και να συμμορφωθούν με αυτό. Άλλα προβλήματα με το πρωτόκολλο προέρχονται από τη διαπραγμάτευση που θεωρούμε ότι, θεωρείται ότι δεν ήταν απόλυτα ορθή και τέλεια όταν γίνεται διαπραγμάτευση δυνατοτήτων αλληλεία σε σχέση με διάφορες κατηγο... διαφορετικές κατηγορίες και διάφορα τμήματα του στόλου, πρέπει και τα τεχνικά μέτρα να διαπραγματευόμαστε κάθε φορά. Δεν έχει ε, νόημα να εκπονούμε συμφωνίες ε, για δυνατότητες αλληλείας όταν τα τεχνικά μέτρα δεν αντιστοιχούν με αυτά. Και εδώ υπήρξαν προβλήματα σε σχέση με τη διαπραγμάτευση που μετά μέσω της Μικτής Επιτροπής ε, ποτέ δεν επιλύθηκαν. Και τελευταίο είναι το θέμα της τομεακής υποστήριξης ε, και που αναμίχθηκε αυτό με τα άλλα θέματα και πραγματικά εδώ υπάρχει πρόβλημα χρήσης των κονδυλίων όσον αφορά την τομεακή ανάπτυξη της αλληλείας ε, στη χώρα αυτή. Όλα αυτά προσωπικά πιστεύω ότι οφείλονται στο ότι δεν είχε η Μαυριτανία μια αυθεντική πολιτική αλληλείας ε, και αν δεν υπάρχει μια αυθεντική πολιτική αλλίας, δεν γνωρίζουν ποια είναι, ποιοι είναι οι στόχοι βραχυπρόθεσμα ε, και μακροπρόθεσμα και δημιουργούνται δυσκολίες και όσον αφορά και την τομεακή ανάπτυξη αυτού του τομέα από πλευρά του. Μας διασφάλισαν όμω ότι σε ένα εγγύς μέλλον θα είναι πρόθυμοι να τα επιλύσουν αυτά και να τα ρυθμίσουν. Σήμερα δεν έχουν ακόμα επιληθεί. κυρίω ο Υπουργό Οικονομικών είπε ότι ο ίδιος θα εγγυόταν ότι στο μέλλον θα συμμορφωνόντουσαν και θα υλοποιούσαν όλες τις προϋποθέσεις ώστε τα κονδύλια να στοχεύσουν στην τομεακή ανάπτυξη. από Α, βγήκε ο κύριος Καντέκα. <clears throat> Αν κάποιος θέλει να προσθέσει κάτι πέρα από αυτά που είπα εγώ και εκτός αυτών οι σχέσεις με τις αρχές ε, όλα αυτά αναπτύχθηκαν σε ένα θετικό πλαίσιο. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημεία που θεωρώ ότι είναι τα ουσιοδέστερα και που έπρεπε να σας αναφέρω από τις ε, συναντήσεις και συζητήσεις που είχαμε. Εν πάση περιπτώσει η γραμματεία έκανε και ένα σημείο, μας συνέταξε και είναι και οι προσωπικές μου αυτές ε, θέσεις. Θα ήθελα να ξέρετε τι γίνεται με την αντιπροσωπεία. Ζητήσατε εσείς τον λόγο, παρακαλώ. Ναι, ε, όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, όταν έχετε μια συνάντηση με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, αν δεν είναι ε, μυστικό, μπορείτε να μας πείτε κάτι για το θέμα αυτό. όταν πήγαμε μας ε, ανακοίνωσαν ότι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης ήθελε να συναντήσει την Ευρωσοπία. Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε μαζί του, αλλά και με οτιδήποτε άλλο. Να πω ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Μαυριτανία είναι ένας, ε, μια, ένας θεσμός ε, αναγνωρισμένος ε, από την πολιτεία. Δεν θυμάμαι, υπάρχουν 50 ή 60 κόμματα στην αντιπολίτευση και αυτός είναι ο ηγέτης και ο πρόεδρος όλων αυτών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Προέρχεται από ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, δεν θυμάμαι το όνομά του, εμπεστώσει είναι ενταγμένος στην ε, σοσιαλιστική διεθνή. Και εξέφρασε την απογοήτευσή του που δεν υπήρχε ε, στην επισοπία μας κανένας σοσιαλιστής. Ε, είπαμε ότι ήμασταν ανοιχτοί, αλλά κανένας σοσιαλιστής δεν ε, αποφάσισε να συμμετάσχει στην ευρωσοπία αυτή. Και επίσης μας εξέφρασε τις ανησυχίες του για τις νέες διαπραγματεύσεις, όπως ε, και για την ε, συμφωνία η οποία συμφωνία θα έπρεπε να είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, να αφορά στην αηφόρο ανάπτυξη, ανησύχησε, ανησύχησε πολύ, απέτεινε κάποιες, ε, έκανε μάλλον κάποιες ερωτήσεις για την ε, παράνομη και ανεξέλεγκτη αλληλεία. Να πω ότι ο κύριος Ισκένο, ε, κάπως έτσι δεν, δεν καταφέρνω να το προφέρω το όνομά του. Ο κύριος ε, αυτό λοιπόν συνοδευόταν από διάφορους ε, βουλευτές της πολιτικής του ομάδας που με με λίγα λόγια εξέφρασαν τις ανησυχίες τους αναφορικά με τις νέες διαπραγματεύσεις αλλά και για το γεγονός πως η η νέα συμφωνία θα έπρεπε να αφορά την αηφόρο ανάπτυξη και την ε, πλά, την παράνομη και ελαφραία αλία. Επίσης δήθηκε το θέμα των επενδύσεων που θα πρέπει να κάνουμε εμεί ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην χώρα, ιδιαίτερα στον τομέα των αλληλευτικών στόλων και τονίσαμε την σημασία της ε, ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών, διότι αν έχει υποδομών δεν μπορεί να επενδύσει ο κλάδος ε, ε, σε αλληλευτικό στόλο. Έχει, είναι, πρόκειται για ένα κρότος το οποίο προσφέρει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, των εξορυκτικές ε, δραστηριότητες όπως πετρέλαιο κλπ. Όπως σα είπα το 30% των εσόδων της χώρας προέρχονται από την Αλία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι σημαντικό για αυτού να διατηρηθεί η συμφωνία προκειμένου να δέχονται αυτές τις ε, μεταφορές ε, χρημάτων Ευχαριστώ τους τρεις ε, βουλευτές που έμειναν μέχρι τελευταία στιγμή εδώ. Πραγματικά είναι λυπηρό να προεδρεύεις επιτροπής όπου ελάχιστοι βουλευτές προσέρχονται. Εν πάση τι να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε στις 3 με την ακρόαση που έχουμε για τις γυναίκες και ελπίζω να έρθει και κάποιος άντρας, να με αφήσουν μόνη μου, διότι ε, εξάλλου αυτό ήταν και αίτημα της ε, σοσιαλιστικής ομάδας. Ευαισθητώς έχω κουραστεί να κάθομαι εδώ και να μην μπορώ να μετακινηθώ. πρόεδρε, ευχαριστεί τους διερμηνείς και εμείς ευχαριστούμε την πρόεδρο. Διακόπτουμε τις μέχρι τις 15.00.